Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω όλους θερμότατα, όλους εσάς τα πλήθη εδώ πέρα που ήρθατε αλλά όλος ιδιαιτέρως να καλωσορίσω τους παρόντες. Κρίμα για την παρουσία. Αύριο θα το λυπηθούν, θα το μετανιώσουν που χάσανε αυτοί. Πρέπει να πάρουμε πρώτα μια σημαντική απόφαση και μετά να συζητήσουμε σημαντικά θέματα. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Δύο υποδείξεις μόνο. Στις συνεδρίες των συντονιστών συζητήσαμε και αποφασίσαμε να δώσουμε μερικές εκθέσεις μπορείτε να τα διαβάσετε στα αντίστοιχα πρακτικά της συνεδρίας αυτής και επίσης συζητήσαμε το θέμα κάποιων προτάσεων που έγιναν για μελέτες, αντιπροσωπείες και ακροάσεις για το 2010. Πολύ γενικά ως πρόταση το κάναμε αυτό γιατί θελήσαμε να έχουμε και χρόνο ε, να το δούμε σε λεπτομέρειες και να το διευκρινίσουμε, αλλά επειδή υπήρχε προθεσμία χρειάστηκε στη διάσκεψη των Προέδρων να το υποβάλουμε αυτό. Ελπίζω να ήταν και το σωστό όργανο η διάσκεψη των Πρόεδρων. <laughs> Δεν ξέρω ποια είναι η αρμοδιότητα εκεί. Υποθέτω ότι συμφωνείτε με αυτά που σας λέγω και περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι η επίσκεψη του κυρίου Ρολσέν και Γενικού Διευθυντή του, Γενικού, του Κοινού συγγνώμη, Κέντρου Ερευνών που παρουσιάζει το θέμα μιας μελέτης και θα έχει και την ευκαιρία συζητήσει μαζί μας. Είχε την καλοσύνη να ε, έχει αυτή την προθυμία. Σας ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζετε όλοι οι παρόντες ότι είναι σημαντικό το κοινό κέντρο έρευνών του οποίου προείσταται ο κύριος Σέγκελ, το θέμα πώς θα αναπτυχθεί στο μέλλον η Ευρώπη, πάρα πολύ σημαντικό, τι θα κάνουμε στην έρευνα και στην καινοτομία. Ε, το έχουμε συζητήσει άλλωστε αυτό το θέμα επανειλημμένα. Είχαμε και κριτικές, ε, επικριτικές ερωτήσεις. Το καλύτερο είναι να τα συζητάμε με τον άμεσα ενδιαφερόμενο και το πιο ευφυές. Και τι να κάνουμε, όποιο έχασε αυτή την ευκαιρία, έχασε, δεν θα την ξαναβρει. Κύριε Σέγκερ, χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Θέλω να σας δώσω το λόγο. Ή δεν είναι πρώτη φορά που έρχεστε εδώ για να μας ενημερώσετε, είναι επανειλημμένα και ούτε και το τελευταίο ραντεβού μας είναι. Αυτό το λέω απειλητικά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Α, θα μιλήσω αγγλικά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι για την ευκαιρία που έχω να σας παρουσιάσω το έργο μας αυτό τον καιρό και προς τα πού κινούμαστε για το μέλλον. Αυτό θα είναι το βασικό τμήμα της παρουσίασης που θα σας κάνω σήμερα. Θα προσπαθήσω μέσα σε 20-25 λεπτά να σας τα παρουσιάσω, παρόλο που υπάρχουν πολλές διαφάνειες. Πάμε στην επόμενη. Θέλω να σας δώσω μερικά παραδείγματα ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και πού βαδίζουμε προς τα πού πηγαίνουμε στο μέλλον. Καταρχήν ποια είναι η αποστολή μας. Εμείς θεωρούμε τον εαυτό μας υπηρεσία της Κομισιόν για να δώσουμε επιστημονικά τεκμηρωμένη συμβολή σε αυτούς που χαράζουν πολιτική. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ αυτό και τι εργαλεία έχουμε. Από τότε που μας δόθηκε αυτή η αποστολή και έχουμε αυτή την δήλωση αποστολής, η υπηρεσία μας ενισχύθηκε και έχουμε εστιαστεί σε αποτελέσματα. Είμαστε κάπως μοναδικοί στην Κομισιόν με την έννοια ότι είμαστε η μόνη γενική διεύθυνση που έχουμε διοικητικό συμβούλιο από τα κράτη-μέλη. Και δεν μας δίνουν μόνο στρατηγική συμβουλή. Παίρνουν μέρος και στον διορισμό των ανώτατων στελεχών της διοίκησης. Μόνο σε εμάς συμβαίνει αυτό. Έχουμε και ένα ε, υψηλό επίπεδο ομάδα χρηστών στην Ένωση, άρα η έγκριση γίνεται και από τα κράτη-μέλη και από τους κύριους πελάτες μας στην Κομισιόν. Και έχουμε και ένα, μια ομάδα interface με τεχνιακή ας συνεργασία δηλαδή με το Κοινοβούλιο. Θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Επόμενη διαφάνεια. Έχουμε 7 Ινστιτούτα σε 5 κράτη-μέλη. Ένα για υλικά ε, αναφορών και μέτρων στο Γκέλ στο Βέλγιο, στο Βορρά. Ένα κέντρο Ινστιτούτο για την Πυρηνική Ενέργεια στην Καλσρουέ, το Ινστιτούτο για την Ενέργεια στην Ολλανδία, στο Βορρά, μια ώρα πάνω από το Άμστερνταμ, τρία Ινστιτούτα στην Ιταλία, ένα στο Ίσπρα, προστασία και ασφάλεια του πολίτη, περιβάλλον και βιωσιμότητα ε, υγιεινή και προστασία του κατανοητή. Και άλλο ένα Ινστιτούτο στην Ισπανία, στη Σεβίλη, για τεχνολογικές μελέτες του μέλλοντος. Και αυτοί κατά κάποιο τρόπο θα αποτελέσουν το κέντρο για υπηρεσίες της Ένωσης σε θέματα περιβάλλοντος, αλλαγής του κλίματος, γεωργίας κλπ. Τώρα, τι ακριβώς κάνουμε. Το πιο σημαντικό προϊόν είναι υποστήριξη σε πολιτική που να στηρίζεται στην επιστήμη. Έχουμε κάμποσα εργαλεία, θα επανέλθω σε αυτό στο τέλος. Δεύτερη δραστηριότητά μας είναι η λειτουργική υποστήριξη, operational support, στην καθημερινή δουλειά. Προβλέπουμε ορισμένα που θα συμβούν, ειδοποιούμε όταν χρειάζεται, παραδείγματο χάρη για την κρίση για τον έμπολα, για τη γρήπη, σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπου μπορεί να εμφανιστεί κάποιο κρούσμα που μπορεί αργότερα να αποτελέσει κίνδυνο, σοβαρό κίνδυνο για τον πολίτη. Αντιμετώπιση των κρίσεων, α το πούμε, η πρόληψη των κρίσεων. Διαχείριση των κρίσεων. Τρίτη δραστηριότητα, είμαστε ένα κέντρο αναφορά, επιστημονικό και τεχνικό το επόμενο slide. Συμμετέχουμε σε όλο τον κύκλο της πολιτικής. Εκεί που είμαστε σχετικά ασθενείς, τολμάω να το πω, είναι στη, στην, στις προβλέψεις, πρόορες κινήσεις. Τι νέες εξελίξεις θα έχουμε στην επιστήμη που μπορούν να έχουν, να να έχουν κάποιον κίνδυνο για τον πολίτη. Και εκεί αυτός που χαράζει την πολιτική θα πρέπει να αντιδράσει έγκαιρα για να προλάβει τον κίνδυνο. Και ένα δεύτερο ασθενέ σημείο είναι η αξιολόγηση εκ των υστέρων, ex post. Πάρθηκε μια απόφαση, πρέπει μετά, εκ των υστέρων δηλαδή, να γίνει μια αξιολόγηση. Το πέτυχε η πολιτική αυτό που ήθελε να κάνει ή όχι. Επόμενο slide. Κατανομή του προπολογισμού. Το πιο μεγάλο κομμάτι είναι η υποστήριξη της ευημερία. Πολιτική χημικών, βιοτεχνολογία, ενέργεια, μεταφορές, κοινωνία της πληροφορίας. Μετά έχουμε αυτό που λέμε δράσεις αλληλεγγύης, περιβάλλον, κλίμα, ανάπτυξη της υπαίθρου. Μετά είναι το πυρηνικό μας πρόγραμμα, ιδιαίτερα σε θέματα ασφάλειας εσωτερικής και εξωτερικής. Και τέλος η, η ασφάλεια από εξωτερικούς κινδύνους. Επόμενο. Μερικά παραδείγματα του τι κάνουμε. Υποστηρίζουμε τη Γενική Διάθεση Τρέν στα σχέδια ε, στρατηγικής τεχνολογίας για την ενέργεια. Χάρτες της ενέργειας, χάρτες δυναμικού, πυρηνική ασφάλεια, απόδοση των διαφόρων μονάδων παραγωγής και τρόπων παραγωγής και έρευνα για τα φωτοβολταϊκά κύτταρα Επόμενο slide. Εδώ έχετε λεπτομέρειες. Απλώς είναι ένα παράδειγμα. Μιλάτε για τα βιοκαύσιμα. Weld wheels όπως το λέμε. Πρέπει να ε, δώσουμε πιστοποιητικά του 60% όλων των ε, κομματιών, των φωτοβολταϊκών κομματιών και σχημάτων που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Γιατί το κάνουμε αυτό. Πολλοί λένε ότι η αποδοτική ε, όσον αφορά τα νούμερα τη απόδοση είναι άριστα. Ωστόσο αν πάει κανεί στο εργαστήριο και συγκρίνει βλέπει ότι αυτό ο ισχυρισμό δεν στέκεται πάντα. Εμεί λοιπόν είμαστε ένα εργαστήριο πιστοποίηση. Ελέγχουμε ότι αυτά που ισχυρίζονται διάφορα και κλπ. είναι σωστά. Άλλη διαφάνεια. Κλιματολογικές αλλαγέ. Εμεί δημιουργούμε μοντέλα. Στην πρώτη πρόταση πριν από δύο χρόνια αναλύσαμε το σενάριο business as usual. Ότι τάχα δεν θα αλλάξει τίποτα. Τι εξελίξει θα έχουμε τα αέρια θερμοκηπίου και μετά κάναμε άλλα μοντέλα τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλον. Αν θέλουμε να περιορίσουμε κατά τόσου βαθμού, τι πρέπει να κάνουμε και πώ για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Άλλο, άλλη διαφάνεια για την αλληλεπίδραση που υπάρχουν ανάμεσα στα διάφορα μοντέλα και σύνολα δεδομένων για τις κλιματολογικές αλλαγές. Έχουμε όλα τα μοντέλα για να κάνουμε σενάρια καθολικά όσον αφορά την ενέργεια. Όπως επίσης έχουμε και σχήματα που μας επιτρέπουν να μπούμε στις βάσεις δεδομένων, δούμε τι εκπομπές και τι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έχουμε από ρηπαντές. Τρέχουμε αυτά τα μοντέλα και βλέπουμε τι αποτέλεσμα μας δίνουν για τη ρήπανση στον αέρα, ε, η χημεία πώς επηρεάζει την ατμόσφαιρα, το έδαφος, οι που πώς επηρεάζουν και προσπαθούμε να υπολογίσουμε ποια θα είναι η επίπτωση στην αλλαγή, της αλλαγής του κλίματος στην υγεία, στη γεωργία, στην οικονομία. Υποστηρίζουμε τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλον και άλλες γενικές διευθύνσεις. Επόμενη διαφάνεια. Με μικρά γράμματα. Σας είπα πώς αντιδρούμε σε κρίσεις. Τα τελευταία δύο χρόνια βλέπετε εδώ πολλά παραδείγματα για το σεισμό στο Αμπρούτσο στην Ιταλία, μια αξιολόγηση των ζημιών και παρακολουθούμε το θέμα. Συχνά όταν υπάρχει μια σοβαρή καταστροφή, που όμως χάρη πυρκαγιές δασών ή σεισμοί, κάποιος δεν το λόγο. Όχι, συνεχίστε, εμείς σημειώνουμε τα ονόματα. Όταν έχουμε μια τέτοια κρίση, εμείς υποστηρίζουμε τους πελάτες μας προκειμένου να κάνουμε μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της ζημιάς, γιατί οι χώρες μας να ζητήσουν να χρησιμοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ένωσης. Εμείς πρέπει να ελέγξουμε ότι το νούμερο ανταποκρίνεται στις, στην πραγματική ζημιά. Επόμενη διαφάνεια. Μέχρι επόμενη διαφάνεια και εδώ έχουμε παραδείγματα πώς βοηθάμε την έρευνα στο ERA Watch και στα δίκτυα ERA αυτό με τη Γενική διάθεση Έρευνας. Δεν βλέπουμε τις πληροφορίες που υπάρχουν, τις εξελίξεις που υπάρχουν στα κράτη-μέλη και σε περιφέρειες και από κοινού ετοιμάζουμε μια έκθεση αναλυτική κατά χώρα με δείκτες προκειμένου να έχουμε πληροφορίες και δεδομένα που θα μας βοηθήσουν να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην έρευνα στην Ένωση. Επόμενη διαφάνεια. Αυτό είναι το scoreboard όπως το λέμε που το δημοσιεύεται κάθε χρόνο. Συλλέγουμε στοιχεία από επενδύσεις σε όλο τον κόσμο. Από εταιρείε, από τον ιδιωτικό τομέα δηλαδή, παρακολουθούμε τις, πιο μεγάλες, τις χίλιες πιο μεγάλες βιομηχανίες στην Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες περιοχές και συγκρίνουμε τα στοιχεία αυτά επενδύσεων για να διδαχθούμε. Και κάνουμε μια ανάλυση της κατάστασης, τι γίνεται στην Ευρώπη και τι γίνεται με τις άλλες χώρες στον κόσμο. Τι δίνει η σύγκριση. Η πρόσφατη αυτό, πίνακας αυτός ε, των μετρήσεων μας δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επενδύονται πάρα πολύ. 8 με 9% είναι μέση επένδυση στην Ένωση. Αρκετά ψηλή ω νούμερο σε σύγκριση με τις ΗΠΑ. Ωστόσο υπάρχει μια διαφορά, ιδιαίτερα στον αφορά στη βιομηχανία υψηλή τεχνολογίας. Επόμενη διαφάνεια. Γάμα μειόμικρον γενετικά μεταλλαγμένα. Εμεί είμαστε το εργαστήριο τη Ένωση. Συντονίζουμε τη δουλειά όλων των εργαστηριών. Και βλέπουμε κατά πόσον συμμορφώνονται αυτά τα προϊόντα σε σχέση με του κανόνε εμπορία του. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να έχουμε στρεβλώσει στο εμπόριο τα επόμενα χρόνια, διότι έχουμε 30 γενετικά μεταλλαγμένα προϊόντα στην Ένωση αυτή τη στιγμή, αλλά σε τέσσερα χρόνια από 30 θα γίνουν 120 γάμα μειόμικρον. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις εγκρίσει προκειμένου να εφαρμόζονται ομοιογενώς σε όλη την Ένωση. Επόμενη διαφάνεια. Βοηθάμε και στην έρευνα δίνοντας πρόσβαση σε σημαντικές υποδομές. Σας είπα ότι είμαστε εργαστήριο αναφορά ανταλλαγμένα. Αλλά έχουμε 7 τέτοια εργαστήρια αναφοράς όπου παίζουμε διαιτητικό ρόλο για τις εκπομπές υποδομές γενικά όπου και έρευνα κάνουμε και δίνουμε πρόσβαση σε ερευνητές από όλο τον κόσμο και εκπαιδεύουμε. φοιτητές μεταπτυχιακά και άτομα από υποψήφιε χώρε που υποφελούνται και αυτέ από την εμπειρία μα. Η επόμενη διαφάνεια είναι πολύ πλοκό, θα μπορούσαμε να το περάσουμε γιατί ουσιαστικά μιλάμε για ένα δίκτυο αριστείας που υπάρχει που το συντονίζουμε με τρία άλλα μεγάλα εργαστήρια στην Ένωση προχωρούμε τα διεθνή πάνελ υπό τον ε, David King. Έγινε μια αναθεώρηση από τους ε, ειδικού εμπειρογνώμονες πέρυσι με θεωρητικά πορίσματα λένε ότι είναι πεπισμένη για την άρεστη ποιότητα στο έργο και τις πολιτικές που υποστηρίζουμε αλλά ένα σωστό πάνελ και είναι στο πάνελ, πρέπει να κάνει και συστάσεις χρήσιμες και τις εφαρμόζουμε. Μία είναι να δρούμε πιο γρήγορα, πιο έγκαιρα, να είμαστε πιο προδραστικοί. Είναι μια σύσταση προς την Κομισιόν αυτή. Προχωρούμε. Εδώ είναι σημαντικό για μας το να έχουμε, να κρατήσουμε ψηλά την επιστημονική αριστεία και όχι μόνο να μιλάμε, αλλά και να το εφαρμόζουμε. Έχουμε άριστα δημοσιεύματα στο Science, στο Nature και σε άλλους επίπεδα. Έχουμε αιτήσει τελετές απονομής βραβείων για καλές επιδόσεις των συνεργατών μας. Προχωρούμε. Συστάσεις από το πάνελ του David King να έχουμε μια ειδική στρατηγική επιχειρήσεων για τα επόμενα πέντε χρόνια. Θέλουμε να υπάρχει η δυνατότητα πολλών επιλογών για την επιστήμη, διότι από εκεί προερχόμαστε κι εμείς, από τις θετικές επιστήμες. Αλλά δεν έχουμε επενδύσει αρκετά ως τώρα στο επιπτώσεις στην οικονομία, στο περιβάλλον, στην κοινωνία, που είναι σημαντικό για αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Ε, λοιπόν, προσθέτουμε αυτές τις παραμέτρους, αυτές τις αρμοδιότητες, ας το πούμε. Αυτά μας δείχνει αυτή η διαφάνεια. Να έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες και περισσότερο προσωπικό. Υπάρχουν και άλλοι στόχοι στην επόμενη διαφάνεια. Από τη στιγμή που θα έχουν οριστεί η στρατηγική στόχοι από τη στιγμή που θα έχουμε επαφή και συμβουλέ από όλου του πελάτε μα στην Κομισιόν, έχουμε την πρώτη συνάντηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και με την ομάδα εργασία που έχουμε το Κοινοβούλιο, θα τα συζητήσουμε έτσι ώστε από όλε τι πλευρέ να έχουμε ε, εισρωή πληροφοριών και στοιχείων για το τι θα κάνουμε τα επόμενα 10 χρόνια. Πηδάμε ένα slide και πάμε στο επόμενο. τι έχουμε να κάνουμε εμείς από κοινού, με το κοινοβούλιο δηλαδή. Ξεκινώντας το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, η ιδέα της ομάδας εργασίας Ευρωκοινοβούλιο και το ΚΚΕ συναισθήθη, διότι εσείς θεωρήσατε ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα ωφεληθεί από τις ε, επιστημονικές γνώσεις του ΚΚΕ. Το κάναμε αυτό, κάναμε μελέτες στη αιτήση του Ευρωκοινοβουλίου επόμενη διαφάνεια βλέπετε τι κάνουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχήν σας πληροφορούμε ποιες είναι οι πρόσφατες εξελίξεις. Ξέρετε τι κάνουμε. δεν να υποστηρίξουμε την Κομισιόν. Περιβάλλον, γεωργία, επιχειρήσεις κλπ. Πού διαμορφώνουμε πολιτική ή που παρακολουθούμε πως εφαρμόζεται η πολιτική είναι ένα φόρουμ όπου οι ευρωβουλευτές και οι επιστήμονές μας έχουν ένα παρεδώσε και αν χρειαστεί σας δίνουμε και επιπλέον πληροφορίες. Επόμενη διαφάνεια, μία μελέτη, για, ε, ένα παράδειγμα μάλλον μελετών που κάναμε για σας. Ένα για την επίπτωση της υγείας στην υγεία των γενικά μεταλλαγμένων τρόφιμα και ζωοτροφές, περισσνό, άλλο για τη βιώσιμη γεωργία και την προστασία του εδάφους, άλλο για προστασία των χημικών που υπάρχουν στον αέρα σε εσωτερικούς χώρους και την κίνηση είναι αυτό για τη υγεία και διάφορες ευκαιρίες προσφέρει η σύγχρονη βιοτεχνολογία. Επόμενη διαφάνεια. Βλέπετε πώς λειτουργεί αυτή η μεταχμιακή ομάδα, η interface. Ο προηγούμενος πρόεδρος ήταν ο Ράινο Πασιλίνα Βλέπετε τι, κάνουμε για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ε, επίπτωση των γενετικά μεταγραμμένων στην υγεία, ένα σημαντικό γραφείο ελέγχου για, τις, για τη ρήπανση και την πρόληψη. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις εκπομπές από τα εργοστάσια στην Ένωση, κλιματολογικές αλλαγές και αυτές. Αυτά παραδείγματα ναι. Και σχεδόν τελείωσα. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι βασικός εταίρος του ΚΚΕ και θέλουμε την αλληλεπίδραση και αμοιβαία δουλειά μεταξύ μας και γι' αυτό ε, ε, ήρθαμε σχετικά νωρίς τώρα στην Επιτροπή σας για όσους δεν ξέρετε να έχετε την ευκαιρία να έχουμε μια επαφή και η τελευταία διαφάνεια στις 28 Οκτωβρίου θα έχουμε την, τα εγγένεια κατά κάποιο τρόπο της πρώτης ετήσιας διάλεξης στις Βρυξέλλες. Πάρα πολλά άτομα έχουν γραφεί να μιλήσουν. Ο μιλητής είναι ο από την Αμερικανική Ένωση για την Πρόθεση της Επιστήμης, ο Άλαν Λέσνερ, ο επικεφαλής. Αυτός είναι επικεφαλής, είναι ο, ο το υπαριθμόν ένα πρόσωπο στην Ένωση αυτή και θα μας μιλήσει για τη συνεργασία Ευρώπη-Αμερική. Και τον Μάιο του χρόνου θα γίνει μια έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο 3 με 6 Μαΐου όπου θα σας πούμε τι κάνουμε. Αυτά είχα να σας πω μέχρι στιγμής και έχετε την ευκαιρία να κάνετε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γενική Διευθυντά, για την εκτενέστατη αυτή ενημέρωση, πάρα πολλά μας είπατε και ήδη έχουν ζητήσει το λόγο γιατί ξύπνησατε την περιέργεια σε πολλούς συναδέλφους και θέλουν πρώτα να κάνουν ερωτήσεις ή να εκφράσουν απόψεις με τη σειρά. Ποιος ζήτησε πρώτος το λόγο. Η κυρία Γκουτιέρες Κορτίνες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Ανισχώ λίγο πρέπει να σας πω. Διότι ε, παρατηρώ ότι αυτά τα μεγάλα ερευνητικά κέντρα που έχουν πολυπολιτισμική διάσταση και στην έρευνα, ε, δηλαδή διεπιστημονική έρευνα, πολλά τα μέτωπα και θα πρέπει να παρακολουθούν και την πολιτική στην έρευνα. Αλλά Εκεί μου λείπουν δύο πράγματα. Πρώτον, η ευρωπαϊκή τάση να κάνει πάντα διάγνωση, δείκτες, παρατηρήσεις. Πολύ ώρα τα περιγράφουμε. Οι λύσεις που είναι. Η μεγάλη διαφορά σε ένα μεγάλο τμήμα της έρευνας που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό που κάνουν ορισμένα κέντρα ερευνών εδώ είναι ε, εκεί κοιτάνε ποιες είναι οι λύσεις στα προβλήματα. Πολύ ωραίοι οι χάρτες. Με, με εκτός από τους χάρτες, καμιά λύση έχουμε. Γιατί ο χάρτης παντού το περιγράφει ίδιο το πρόβλημα, αλλά τα προβλήματα δεν είναι παρόμοια. Ας πούμε, ε, τα προβλήματα στις κατολιστήσεις ε, ή στο έδαφο δεν είναι τα ίδια στη Σικελία ας πούμε, και στη Βόρεια Ευρώπη. Είδατε τι έγινε στη Σικελία πρόσφατα. Δεν είναι ίδια η λύση αλλού. Και εσείς μιλήσατε για άλλους τομείς. Εγώ θέλω περισσότερη προσπάθεια να γίνεται για τη λύση, για τη θεραπεία, όχι για τη διάγνωση. Καταλαβαίνω ότι το κέντρο αυτό δεν κάνει έρευνα μόνο του, αλλά κάνει συμπιλήματα, συνόψεις και προτείνει πρωτοβουλίες. Λοιπόν, το δεύτερο που ήθελα να πω είναι, ας πούμε, στη γεωργία και στην αηφορία. Αν κοιτάξουμε τι έγινε στο παρελθόν, Θυμάστε τη Μαφάλντα. Η Μαφάλντα αυτό το ε, καρτούν ε, έλεγε ότι κοιτάει το μέλλον με τα μάτια της στο σβέρκο. Εμείς δεν μπορούμε να κοιτάμε το μέλλον με τα μάτια στο σβέρκο. Ε, άλλη παραγωγικότητα είναι σήμερα, άλλα τα προβλήματα σήμερα. Χρειάζεται περισσότερη γεωργία γιατί ε, αυξάνεται ο πληθυσμός του κόσμου και θα πρέπει να τον ταΐσουμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να σκεφτόμαστε ε, τις βραδικίνητες δομές της σημερινής γεωργίας. Τι κάνουμε, έχουμε κλιματική αλλαγή, έχουμε υπερπληθυσμό. Ε, θα πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη έρευνα, ας πούμε, για την έγκαια βελτίωση, για τα ποτίσματα. Το κέντρο σας, λοιπόν, θα πρέπει να κάνει μια προσπάθεια για να εντοπίσει κάποιες αντιφάσεις που ζούμε στην Ευρώπη. Και πραγματικά βάζουμε τρικλοποδιά στον εαυτό μας, πυροβολούμε το πόδι μας, ας πούμε, παράδειγμα. Κοιτάξτε τι λέει τον Αύγουστο το περιοδικό Nature για το πρόγραμμα REACH. Η Ευρώπη πολλαπλασιάζει επί 50 τον αριθμό των αναλύσεων και των ε, μελετών και των πειραμάτων σε ζώα. Τι έλεγε το REACH, να μειωθούν τα πειραματόζωα. Ε, τώρα τι κάνει η Ευρώπη. Θα σας στείλω στους συναδέλφους το άρθρο, είναι πραγματικά ε, εντυπωσιακά αυτά. Μία ιδέα αυτή. Δεύτερο, στην Σουηδία ή στην Νορβηγία νομίζω υπάρχει μια ιδέα που έχει αναπτυχθεί για το ποιες είναι ευρωπαϊκές οδηγίες που βλάπτουν την ιστορική κληρονομιά. Ας πούμε, απαγορεύουμε το μόλιβδο και δεν μπορούμε να, να επισκευάσουμε τα βιτρό στους καθεδρικούς ναούς. Έχουμε κάποια κτίρια ε, ιστορικά και ιστορικές πόλεις και η νομοθεσία μας δεν τα σέβεται και δεν σέβεται τη συντήρησή τους. Άλλο παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει για να ξεπατώνει δέντρα στη Νότια Ευρώπη. Εκρίζωση. Ε, ε, και αμπέλια ξεπατώνονται. Και ε, είναι υπερονόβια δέντρα και το καλύτερο κρασί βγαίνει από τα παλιά αμπέλια που εμείς ξεπατώνουμε. Και εμείς τα πληρώνουμε όλα αυτά. Και αυτό ε, είναι υπέρ της διάβρωση των ε, εδαφών, γιατί δεν συγκρατείται το χώμα και φεύγει. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει μια ειδική έρευνα για το ποια επίπτωση έχει κάθε νομοθέτημα στη φύση μας, γιατί από τη μια ε, σπέρνουμε και από την άλλη ε, ξεπατώνουμε. Ευχαριστώ. Κύριος Κορέρα Ντεκάμπος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον καθηγητή Σέγκελ για την εξαιρετική του παρουσίαση για τις δραστηριότητες του κέντρου και θα ήθελα να πω το εξή. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή η εξέλιξη του Ιδρύματος με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον το υλικό που μας δώσατε είναι και αυτό πολύ ενδιαφέρον και όχι μόνο από ιστορικής άποψης. Έχω την εντύπωση ότι πραγματικά είναι ενδιαφέρον να κάνουμε μια ανάλυση της ιστορικής εξέλιξης του Ιδρύματος γιατί στη τελική ανάλυση αποτελεί μια εξέλιξη η οποία δεν μπορούσαμε να την προβλέψουμε πριν από 20-30 χρόνια. Αναπτύχθηκε μια ξεχωριστή δυναμική και τώρα μόλις τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε η ειδική στρατηγική και διάβασα τα έγγραφά σας. Φαίνεται ότι το κέντρο ασχολείται ουσιαστικά με τα προβλήματα αυτά με οικονομικό τρόπο ή μήπως αυτό είναι κάτι το τυχαίο. Διαπιστώνω ότι αρχικά, για παράδειγμα, τα θέματα πυρηνικής ενέργειας και της ασφάλειας των πρινικών εργοστασίων αποτελούσαν θέματα βασικής ε, σημασίας και αργότερα βλέπω ότι η προσοχή στρέφεται στο soft science, την πιο ήπια επιστήμη και στη συνέχεια αναπτύσσεται μια διαφορετική γραμμή. Διαπιστώνω λοιπόν ότι ε, υπάρχουν διάφοροι ευγενείς ε, σκοποί. Το θέμα είναι έτσι θα μείνουν τα πράγματα. Βάσει της εμπειρίας σας θεωρείτε ότι ποια θα είναι η εξέλιξη, έστω ότι σας δίνουν λευκή επιταγή. Τι θα κάνετε στο μέλλον. Θα προτείνετε ένα νέο διοργανωτικό μοντέλο, θα αντιδρούσατε με διαφορετικό τρόπο στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Πώς θα προτιμάσατε την στρατηγική σας. Ξέρω ότι φυσικά η ο προπολογισμό και οι χρηματοοικονομικέ ε, προοπτικέ ε, σα περιορίζουν και φυσικά μπορεί και εσεί να έχετε ελπίδε για βελτιώσει, αλλά θα δούμε τι θα γίνει σε κάποια χρόνια τελικά. Ευχαριστώ, συνάδελφο Γκίρεκ. E, e, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ έχω μία ερώτηση να απευθύνω προς τον καθηγητή Σέγκελ. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να έχει εντολή για να δράσει σε ό,τι αφορά το πακέτο για το κλίμα. Αλλά για να λάβει την εντολή αυτή, χρησιμοποίησε ένα μοντέλο το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα αξιόπιστο, το οποίο ουσιαστικά ε, κατέληξε σε ένα στόχο, σε ένα θέμα, στις αλλαγές ε, στο διοξείδιο του άνθρακα και στην ατμόσφαιρα. Το ερώτημα λοιπόν που έχω να θέσω είναι το εξής. Στο κέντρο σας ε, εργάζεται σε επί μια πιο συνεκτική, αν θέλετε, στρατηγικής από επιστημονικής πλευράς για να ληφθούν υπόψη και άλλα στοιχεία, όπως οι αλλαγέ ε, ε, στις κινήσεις του ηλίου και άλλοι χιλιάδε παράγοντες που επηρεάζουν. Γιατί επιλέξαμε μόνο τον παράγοντα του διοξιδίου του άνθρακα και θα ξέρετε ασφαλώς ότι με μια ορισμένη μαθηματική, ένας ορισμένος μαθηματικός τύπος μπορεί να χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους ανάλογα με τι παράγοντες θα χρησιμοποιήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια επιστημονικά αξιόπιστη προσέγγιση. Ξέρετε κάτι παραπάνω για ένα τέτοιο μοντέλο. Είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ο κύριος Οντί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με τη σειρά μου και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το Γενικό Διευθυντή και συγχαρητήρια κύριε Γενική Διευθυντά για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να σας μεταφέρω μια ανησυχία των βουλευτών. Διότι εμείς εκπροσωπούμε τους πολίτες και ερευνητικούς οργανισμούς με τους οποίους έχουμε επαφές είτε αυτό είναι τώρα δημόσια κέντρα, ιδιωτικά κέντρα, εθνικά κέντρα ερευνών, ανησυχούν και εκείνοι για την εξέλιξη που παίρνουν τα πράγματα. Και δεν είναι καινούριο αυτό άλλωστε. Προετοιμάζοντας τη σημερινή συνεδρίαση, ε, κοίταζα τι έλεγε ο Επίτροπος Μπιουσκέν το έτος 2000. Κραυγή αγωνία για την έρευνα και ζητούσε τη δημιουργία ενό ευρωπαϊκού χώρου Έρευνα. Εσεί είπατε ότι παίζετε ρόλο συμβουλευτικό. Θα μπορούσατε παρακαλώ να διαδραματίσετε αυτό το ρόλο και να συμβουλεύσετε και την, την Επιτροπή μας εδώ ε, να μας πείτε τη γνώμη σας για το πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς μια γνήσια πραγματικά ευρωπαϊκή πολιτική έρευνας. Γιατί είναι πολλά τα θεσμικά όργανα και τελικά τρεις συλλογικέ σε αυτό το τόσο περίπλοκο τοπίο της έρευνας. Πρώτα έχουμε μια διακρατική λογική, διακυβερνητική οι κυβερνήσεις ε, χειρίζονται τα μέσα, τα κράτη-μέλη δηλαδή. Η δεύτερη λογική είναι διοργανική. Υπάρχουν θεσμικά όργανα, ιδρύματα, Ινστιτούτα και συνεργάζονται μεταξύ τους. Και το τρίτο είναι αυτό που κάνουμε εμείς σε κοινοτικό επίπεδο. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό τον κικαιώνα, πώς θα μπορούσαμε πώς να, το να βρούμε μια συνοχή μια ευρωπαϊκή πραγματικά πολιτική έρευνα. Και έρχομαι στη δεύτερη ερώτησή μου που είναι η χρηματοδότηση. Σήμερα 80% περίπου της έρευνας, αν δεν απατώμε, χρηματοδοτείται από τα κράτη-μέλη. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Γίνεται στα κράτη-μέλη τα ίδια. Πώς μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε χωρίς να αυξήσουμε τους δημοσίους πόρους για να κοινοτικοποιήσουμε περισσότερο τη χρηματοδότηση της έρευνας, όπως κάναμε με τη Γεωργία περίπου. Κατά την άποψή σας αυτό είναι εφικτό, είναι επιθυμητό, είναι πιθανό. Και επίσης έχετε και καλή σχέση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ε, θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο εργαλείο και μπορεί μέσω δανείων να χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα. Πώς το βλέπετε. Γενικά θα ήθελα να σας μεταφέρω μια ανησυχία έτσι, των βουλευτών γιατί δυσκολευόμαστε πολύ να βρούμε τις δομές. Έχουμε και τον Επίτροπό μας που και αυτός ο άνθρωπος ό,τι μπορεί κάνει. Αλλά εσείς ως διευθυντής ενός Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Οργανισμού τι άποψη έχετε για την εξέλιξη της έρευνας για να μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε στον παγκόσμιο ανταγωνισμό αποτελέσματα. Κάποιος ε, έλεγε, ο στρατηγός Δεγκόλ έλεγε ότι έχουμε ερευνητές, αλλά δεν έχουμε ανθρώπους που ψάχνουν δηλαδή, αλλά δεν έχουμε ανθρώπους που βρίσκουν. Ευρώντες, λοιπόν, τι μπορείτε να μας ε, συμβουλεύσετε. Η κυρία ε, Ριέρα Μαντουρέλ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Σέγκελ για την παρουσία σας και την παρουσίασή σας εδώ. Όπως πάντα ήταν πάρα πολύ διαφωτιστικά αυτά που μας είπατε ε, για μας όλους, αλλά όπως είπατε και εσείς πολύ καλά και για τα νέα μέλη, τους νέους βουλευτές που σας βλέπουν για πρώτη φορά. Διότι σίγουρα είναι σημαντική δουλειά αυτή που γίνεται στο κοινό κέντρο ερευνών, αλλά πολλές φορές είναι ο μέγας άγνωστος και για ε, πολλούς Ευρωπαίους και για πολλούς βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μας παρουσιάσετε ωραία τη δουλειά που κάνετε και είμαι πεπισμένη ότι αυτό είναι αλήθεια. Αλλά υποθέτω επίσης ότι και στην καθημερινή σας ζωή δεν είναι τα πάντα εύκολα. Γι' αυτό θα ήθελα λίγο να μας ενημερώσετε για την άλλη πλευρά του νομίσματος. Δηλαδή, θα ήθελα να σας ρωτήσω, Ποιες είναι οι δυσκολίες που έχει ακόμα να αντιμετωπίσει το κοινό κέντρο ερευνών στην καθημερινή του δουλειά. Και αν ανταποκρίνεται στους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε, που είναι η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η υποστήριξή της για τις πολιτικές αποφάσεις. Είναι ανεξαρτησία, η χρηματοδότηση θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι τα μεγαλύτερα ατού σας. Και μετά, πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Έχετε προγραμματίσει ήδη ακόμα και αρχίσει κάτι για το νέο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ε, Έρευνας και Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Έχετε κάποια σχέση εσείς με όλο αυτό. Και σε σχέση με τα όσα ρώτησε και ο κύριος Οντί, μας μιλήσατε για την επιστημονική πολιτική της Ένωσης, αλλά αναφερθήκατε περισσότερο στη σύνδεση της βιομηχανίας των εργοστασίων με τα ερευνητικά κέντρα. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω αν κάνετε τίποτα για τη δημιουργία την ίδια και το σχεδιασμό του ευρωπαϊκού ερευνητικού χώρου. Δηλαδή, κάνετε τέτοιε αναλύσει, ψάχνετε εσεί ποιο θα ήταν ο καλύτερο τρόπο να δημιουργηθεί ο ενιαίο χώρο και η νέα αγορά των ερευνητών. Τι γίνεται με την κινητικότητα των ερευνητών, με τι ερευνητικέ υποδομέ. Σα απασχολεί αυτό ο συντονισμό με τι επιστημονικέ πολιτικέ των κρατών μελών, όλα αυτά. Σα ευχαριστώ πολύ. Αυτέ είναι οι ερωτήσει μου. Ευχαριστώ κύριε ε, Μαντουρέλ. Ο κύριος Μπιτικόφερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Γενική Διευθυντά, σε μία από τις διαφάνειές σας αναφέραστε ότι το, το Κοινό Κέντρο Ερευνών αποτελεί την πιο σημαντική, το πιο σημαντικό ίδρυμα για τους, ευρωπαϊκούς, τους Ευρωπαίους ε, υπεύθυνου ε, για λήψη αποφάσεων σε ό,τι αφορά επιστημονικά τέτοια θέματα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξή. Α υποθέσουμε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν το Συμβούλιο. Και δεν το εννοώ αυτό. Δεν θέλω να κοροϊδέψω το Συμβούλιο. Ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να ζητήσει εθνικούς πόρους. Τι θα γίνει με το Κοινοβούλιο ως φορέα λήψης αποφάσεων. Αυτό που κατάλαβα εγώ για την συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και του κέντρου σας. Δεν ε, κάθεσα το Κοινοβούλιο ως βασικό πάροχο για τέτοια ζητήματα. Πώς θεωρείτε λοιπόν ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να αναπτυχθεί προκειμένου η αποστολή την οποία μας αναφέρατε, η οποία είναι και πάρα πολύ φιλόδοξη παρεπιπτόντως, να αποτελέσει και κάτι το πραγματικό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και χαιρόμαστε που είναι μαζί μας ε, και πάλι ο κύριος Σέγκελ στην Επιτροπή για να μας παρουσιάσει τις δραστηριότητες του κέντρου τις οποίες ε, παρακολουθώ εδώ και αρκετές θητείες. Άκουσα με προσοχή τους συναδέλφους και ανυπομονώ να ακούσω τις απαντήσεις σας. Σε αυτά που ρώτησε ο κύριος Γκέρεκ αναφορικά με τις εναλλακτικέ ε, επιστημονικές έρευνες σε ό,τι αφορά την πολιτική για την αλλαγή του κλίματος. Επίσης, θα ήθελα να ακούσω την απάντηση σε αυτά που ανέφερε ο κύριος Οντή για την κοινή αγροτική πολιτική για την επιστήμη. Δεν κατάλαβα πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό, αλλά θέλω να ακούσω τι έχετε να πείτε κι εσείς και επίσης ε, για την πρόταση, την πρόσκληση του κυρίου Κάμπελ για τα, τα πάνη των πόρων. Φαίνεται ότι εδώ και χρόνια προσπαθούμε να διατηρήσουμε τους πόρους για το κέντρο ερευνών. Δεν είμαι αισιόδοξο για την ε, αύξηση των κονδυλίων, αλλά και πάλι θα ήθελα να ακούσω τι έχετε να πείτε. Το βασικό που θέλω να ρωτήσω ωστόσο είναι το εξή. Θα ήθελα να καλέσω τους συναδέλφους να δράξουν την ευκαιρία για να, επισκέψουν, για να επισκεφτούν ε, ένα και περισσότερα από τα ιδρύματα. Έχω επισκεφτεί αυτό του Σκαλτρούης για παράδειγμα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερα από το να πάτε να δείτε και εσείς ίδια στα μάτια. Και καλωσορίζω την πρωτοβουλία σας να διοργανώνετε εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο εκθέσεις μια έκθεση μάλλον του χρόνου. Μπορεί να έχετε ως επισκέπτες πολλούς από τους βουλευτές στην αρχική σας ομιλία, γιατί είναι και η εβδομάδα τέτοια, αλλά αυτό αποτελεί και ένα πρόβλημα, γιατί γενικά είναι φορτωμένο το πρόγραμμα των βουλευτών. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω τους συναδέλφους να επισκεφθούν τα Ιδρύματα και θα το θέσω το θέμα αυτό και στους συντονιστές της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Τσίθιστερ, θα το συζητήσουμε ίσως ναι και στους συντονιστές μήπως ε, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια προσφορά προς όλη την Επιτροπή. Να βρούμε δηλαδή κάποιο σημείο, μια ημερομηνία για να κοιτάξουμε τα θέματα αυτά. Ο συνάδελφος Βόγκεν. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι η πρώτη φορά που ακούω τέτοια παρουσίαση για το κέντρο και πραγματικά ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Έχω την εντύπωση ότι όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει να υποστηρίξουν το έργο του κέντρου και ιδιαίτερα το έργο που κάνετε για την μελέτη αντικτύπου, γιατί θεωρώ ότι όλες οι πολιτικές μας, όλη η νομοθεσία μας θα πρέπει να εξετάζεται και από αυτή την σκοπιά από τη μελέτη αντικτύπου, δηλαδή με αποδεκτικά στοιχεία. Δεν μίλησατε πολύ για το προσωπικό σας και για τον αριθμό του προσωπικού σας και για την διάρθρωση του, του Ιδρύματος. Το βασικό θέμα της κλιματικής αλλαγής το οποίο έθιξαν και πολλοί συνάδελφοι. Φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά, πολλές ακαδημαϊκές οργανώσεις και επιστημονικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη που αναπτύσσουν τέτοια μοντέλα και υπάρχει και ένα ανάλογο, μοντέλο, ένα ανάλογο ίδρυμα για παράδειγμα στην Βετική Ουαλία. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, με όλες αυτές τις οργανώσεις συνεργάζεστε. Υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, στοιχείων και τη έρευνας, γιατί ασφαλώς με τον τρόπο αυτό δεν θα, θα αποφεύγονταν και οι αλληλεπικαλύψεις. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολλές ερωτήσεις έγιναν. Κύριε Γενική Διευθυντά, κύριε Σέγκελ, έχετε το λόγο και σας επιτρέπουμε να απαντήσετε σε όλα αυτά. Ελπίζω να απαντήσετε τα περισσότερα και αν παραμείνουν ορισμένα ανοιχτά μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις άλλη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ στα αγγλικά η απάντηση. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με τη σειρά που έγιναν οι ερωτήσεις όσο μπορώ. Κυρία Κουτιέρες. Η κυρία Κουτιέρες ρώτησε πολλά ζητήματα και έθεσε και άλλα σωστά και σημαντικά. Θα πρέπει να σας πω όμως ότι ε, το κέντρο μας θα πρέπει να εστιάζει κάπου, θα πρέπει να επιλέγει. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα. Δεν έχω εγώ τη δυνατότητα να σας δώσω όλες τις λεπτομέρειες, αλλά Πρέπει να επιλέγουμε 7-8 μεγάλους τομείς και να εστιάζουμε την προσοχή μας εκεί και να εμένουμε. Δεν ξέρω αν υπήρξε καμία παρεξήγηση να διασκεδαστεί. Εμείς βασικά δουλεύουμε ακριβώ για τις λύσεις. Η διερευνητική έρευνα ή θεμελιώδης έρευνα γίνεται μόνο στο βαθμό που χρειάζεται να αποδείξουμε την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων σε αυτούς τους τομείς κλειδιά. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε ως ρόλο να κάνουμε για καινοτομία ε, η πρωτοπόρα και θεμελιώδη έρευνα υπό τη στενή έννοια και να αφιερώνουμε τα περισσότερα κονδύλια εκεί. Όχι. Το κάνουμε αυτό υποστηρικτικά για να αποδείξουμε ότι οι ερευνητές μας κάνουν εξαιρετική δουλειά, ότι γνωρίζουν αρκετά καλά το πεδίο τους, έτσι ώστε να συνδυάσουν τη γνώση που υπάρχει στην επιστημονική κοινότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για ανάλυση και ε, σεναρίων και ανάπτυξη επιλογών για τις πολιτικές. Αυτή είναι η κύρια απάντησή μου στα ζητήματα που έθεσε η κυρία Γκουτιέρες Κορτίνες. Βεβαίως δεν μπορούμε να καλύψουμε όλους τους τομείς που ανέφερε εκείνη. Δύο λόγια για το άρθρο αυτό στο Nature, για το πρόγραμμα REACH. Ο συντάκτης ήταν πρώην συνεργάτης μας, ήταν επικεφαλής του τμήματος ε, στο Κοινό Κέντρο Ερευνών που ε, εκπώνησε εναλλακτικέ λύσεις προ τι μεθόδους με Μετά πήγε στο Πανεπιστήμιο Τζον Hopkins και ξέρει πολύ καλά ότι ο αριθμός των πειραματοζών που χρειάζεται για το REACH ε, στοιχειοθετείται από διαφορετικά στοιχεία. Και εγώ είχα συγκεντρώσει όλους τους επιστήμονες όταν έγιναν υπολογισμοί για το πόσα πειραματόζωα χρειάζονται για τι διάφορε τοξικολογικέ διάφορες δοκιμές. Και δεν είναι πάρα πολύ θαραλέο να παίρνει κανείς το πια ακραία στοιχεία όταν έχεις μία ψαλίδα, όταν έχεις μία γκάμα. Θα πρέπει ε, να έχουμε ε, ένα αποτέλεσμα που να ευσταθεί και να είναι ισορροπημένο. Πρέπει να σας πω ότι μας έχει δυσαρεστήσει πολύ ε, το άρθρο αυτό και δεν βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία. Τα στοιχεία έχουν χειραγωγηθεί και μεταχειριστεί κάνουν τα στοιχεία αυτά ορισμένοι προς μία κατεύθυνση. Είναι κρίμα για το Nature. Δεν ε, ευσταθούν αυτά που λέει το άρθρο. Ε, για τον κύριο Κορέα ε, Ντεκάμπος, χαίρομαι πάρα πολύ από αυτά που μας είπατε. Γιατί υπάρχει τόσο καλή ανταπόκριση από τους πελάτες μας. Γιατί κάνουμε και μελέτες ικανοποίησης πελατών. Έχω ξεκινήσει και μια σειρά επαφών με όλους τους γενικούς διευθυντές σε τακτικά ε, χρονικά διαστήματα για να κάνουμε και μια ε, πρόβλεψη, ένα χρονικό ορίζοντα, να δούμε τα επόμενα πέντε χρόνια τι αναμένουμε να έρθουν τα αποτελέσματα, ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και πάλι δεν είμαστε μόνοι μας αυτή την προσπάθεια. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών είναι ίσως ο καλύτερος διοργανωτής δικτύων. Έχουμε ε, πολλές εταιρικές σχέσεις και η περισσότερη δουλειά μας γίνεται σε δίκτυα. Σχεδόν καθόλου δεν εργαζόμαστε μόνοι μας, ε, σχεδόν ανέφικτο θα ήταν άλλωστε κάτι τέτοιο. Η πιο δύσκολη ερώτησή σας ήταν πώς θα στήσετε αυτή την οργάνωση, αν θα μπορούσατε να το κάνετε. Είναι πολύ εκανθόδης αυτό το θέμα. Αν θα έπρεπε να το ξανακάνω, δεν θα βάζα ποτέ αυτή τη γεωγραφική κατανομή που έχει γίνει. Είναι σαφώς μειονέκτημα όταν θα πρέπει να έχουμε επιστημονικέ ομάδες που να συνεργάζονται, γιατί αυτό μας χρειάζεται. Είναι σίγουρα μειονέκτημα αυτός ο κατακαιρματισμός που είμαστε σκορπισμένοι σε όλη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα όμως είναι πραγματικότητα. Και τι κάνουμε για να το ξεπεράσουμε, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Τηλεδιασκέψεις πάρα πολύ χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε όλοι μαζί. Και για τις δημοσιονομικές προοπτικές στο σχόλιο σας, η νέα στρατηγική έχει αναπτυχθεί με πρόβλεψη ε, μηδενική αύξηση του προπολογισμού και αυτό είναι η δική μου αντολή. Το είπατε πολύ. Νομίζω θα ήταν λάθος να ζητούσαμε περισσότερα χρήματα. Ίσως δεν θα έπρεπε να βρω έτσι, αλλά έτσι είμαι. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι ε, η διοίκησή μας, τα υψηλόβαθμα στελέχη μας, έτσι σκέφτονται Θέλουμε ε, αναθεώρηση των προτεραιοτήτων, επανεστίαση. Το έχουμε πει και στους πελάτες μας ξεκάθαρα, να επικεντρωθούμε σε ορισμένους τομείς και να μην θελήσουμε περισσότερη ανάπτυξη, μεγέθυνση, ε, αλλά συνεργασία με άλλους σημαντικούς φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον κύριο Γκίρεκ και την κλιματική αλλαγή. Κατά κάποιο τρόπο είμαστε εμείς θύμα των πελατών μας, γιατί λέγεται η στρατηγική μας customer driven, δηλαδή ότι μας ζητάει ο πελάτης που έχει πάντα δίκιο. Και θα πρέπει να σας ομολογήσω ότι έχουμε 70 ή 80 περίπου που εργάζονται στην κλιματική αλλαγή και δεν κάνουμε θεμελιώδη έρευνα. Είναι πραγματικά στην εφαρμοσμένη ε, για στρατηγική ε, περιορισμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και αναπτύσσουμε σενάρια. Το χαρτοφυλάκιο μας λοιπόν εκεί ε, υπαγορεύεται σε μεγάλο βαθμό από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος που είναι ο πελάτης μας και δεν κοιτάμε πολλά άλλα στοιχεία. Εντάξει, παρακολουθούμε όλη τη ιστορία ε, παράλληλα για τη γενετική μηχανική Αλλά πριν αρχίσουμε οποιαδήποτε πειράματα με διάφορα σωματίδια που θα ελευθερώνουμε στο περιβάλλον, χρειάζεται πολύ μεγάλη πληροφόρηση. Γιατί ενδεχομένως οι ε, ζημίες να είναι πολύ μεγαλύτερε από τις ωφέλειε. Λοιπόν, παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά τα θέματα αυτά. Ένας υπάλληλο μα έγραψε και ένα άρθρο για το Science και για το κανάλι του Science για τη γεωμηχανική ε, και τι πιστεύουμε γι' αυτά. Επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Δεν μπαίνουμε σε αυτά τα χωράφια, δεν μπαίνουμε σε βάθος αυτή την έρευνα και δεν θα είχαμε αρρώστα και τη δυνατότητα να το κάνουμε. Επικεντρωνόμαστε στον ανταγωνισμό εμείς σε αυτή την κλιματική αλλαγή και στα οικονομικά στοιχεία για να μπορέσουμε και πάλι να εκτιμήσουμε τις διάφορες μελέτες. Ξέρετε, το Δανό Λόμπαρτ, νομίζω, που μελέτησε τον οικονομικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής. Θέλουμε περισσότερη πραγματογνωμοσύνη εκεί. όχι μόνο τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά, αλλά και τα οικονομικά στοιχεία. Κύριε Οντή, η ερώτησή σας βεβαίως είναι πολύ δύσκολη για μένα. Εμεί δεν κάνουμε ερευνητική πολιτική. Πολλά πράγματα κάνουμε στο κέντρο μα, αλλά όχι ερευνητική πολιτική. Υποστηρίζουμε επιστημονικά ορισμένου τομεί στη Γενική Διεύθυνση Έρευνα, αλλά τον ευρωπαϊκό χώρο, επιστημονικό και χώρο έρευνα κτλ. σε μεγάλο βαθμό το αναλαμβάνει αυτό η Γενική Διεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίω, προσωπικά Πιστεύω ότι για να ενισχυθεί η έρευνα στην Ευρώπη είναι και η κρατική χρηματοδότηση πολύ περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η περισσότερη κρατική έρευνα χρηματοδοτεί ερευνητικά κέντρα στο εσωτερικό των χωρών. Νομίζω θα υπήρχε η υπεραξία εάν τα κράτη-μέλη έδιναν πόρους ή άνοιγαν τα κονδύλια τους ε, στον ανταγωνισμό με κέντρα αριστείας από άλλες χώρες που να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κρατικά κονδύλια των κρατών μελών αλλά με κριτήρια πάντα την αριστεία. Αυτό θα ήταν τεράστιο και υπεραξία και για τα κράτη-μέλη που θα, να μπορούν να χρηματοδοτούν και ε, εξαιρετικές ομάδες ερευνητών από άλλα κράτη-μέλη. Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Γνωρίζω ότι και στην πραγματικότητα όμως πώς έχει η κατάσταση. Η κυρία Ρία Ραμαντουρέλ. Και πάλι σας ευχαριστώ για τα θετικά σας σχόλια. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Νομίζω η μεγαλύτερη μεμονωμένη δυσκολία που έχουμε είναι η συγκέντρωση. Δηλαδή, το περισσότερο προσωπικό απασχολείται, ε, μάλλον, ε, ανησυχεί ε, έχουμε δυσκολίες στην πρόσληψη. Το συζητάμε με την ΕΠΣΟ και με την διοίκηση, τη Γενική Διεύθυνση, την αρμόδια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι βαριές οι διαδικασίες χρονοβόρες. Ε, έχουμε όμως πολύ καλό διάλογο μετά από τις συστάσεις του David King στην έκθεσή του. Χρειαζόμαστε πολύ καλό προσωπικό και θέλουμε να γίνουν ειδικοί διαγωνισμοί για ειδικού ερευνητές που έχουν επιλεγεί πραγματικά για την άριστη επίδοσή τους ε, στην ίδια την επιστήμη και όχι να έχουν κάνει κάπου διαχείριση έρευνα σε διοικητικό επίπεδο. Γι' αυτό έχουμε και μεγάλο βαθμό εκτάκτων υπαλλήλων ε, προβλέψει με ε, επιστημονικούς επισκέπτες, με μεταπτυχιακούς φοιτητές, φοιτητές διδακτορικό που να μετακινούνται και να έρχονται ε, βράχοι πρόθεσμα σε εμά. Τεχνολογία και καινοτομία για το μέλλον σας είπα ήδη ότι έχουμε λάβει ε, απόφαση και συμμετέχουμε σε προγράμματα εφόσον είναι στους τομείς ε, ενδιαφέροντός μας και αρμοδιότητάς μας. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, συμμετέχουμε. Νομίζω ότι για το σχεδιασμό του ΕΡΑ απάντησα προηγουμένως για τον κύριο Μπιούτι Κόφερ είναι απόλυτα σωστό το σχόλιο σας. Καταλαβαίνω τι λέτε. Είχε γίνει μια παρεξήγηση. Έλεγε ο, πιο έμπιστος, ε, the most trusted. Δεν είμαστε ο μοναδικός σύμβουλος. Αυτό θα ήταν άλλωστε αλαζονικό και τελείως ε, ανεδαφικό, αλλά ελπίζω να καταλάβατε από την προηγούμενη μου τοποθέτηση ότι δουλεύουμε ως δίκτυα. Όταν λέμε ε, οι Ευρωπαίοι που φτιάχνουν τις αποφάσεις, κυρίως εννοούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κυρίως έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας. Δηλαδή, ο βασικό μα συνομιλητή και υποστηρικτή είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά τα άλλα, έχουμε μεγάλη διάδραση και με το Κοινοβούλιο. Αλλά ποτέ δεν είπα ότι είμαστε ο μοναδικός, ο μεγαλύτερος ή το μονοπόλιο. Ούτε ποτέ θα ισχυριστώ και θα διεκδικήσω κάτι τέτοιο. Είναι πολύ κακό για το όργανό μας. Δεν θέλω να είμαστε ούτε ο μεγαλύτερος σύμβουλος, ούτε ο μοναδικός. Πρώτον είναι τελείως εθεροβάμων και το δεύτερο είναι πάντα κακό όταν έχεις μονοπόλιο για το ε, κέντρο ερευνών. και με το Συμβούλιο υπάρχει κάποια σχετική συνεργασία για την ασφάλεια, αλλά όπως είπατε τα κράτη-μέλη έχουν ε, ήδη ε, την ερευνητική τους πολιτική σε κρατικό εθνικό επίπεδο, καλά εδρεωμένη και λειτουργούσα και εμείς απλώς συντονίζουμε. Για τον Τσάρλς Τσίτσεστε, προσπάθησα να απαντήσω στο πρώτο σας ε, σκέλος και απάντησα ήδη και στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Δεν ζητάμε επιπλέον χρηματοδότηση, προσπαθούμε να περιοριστούμε στο προϋπολογισμό που έχουμε, αλλά να έχουμε και ανταγωνιστικά έσοδα. Δηλαδή να αποδείξουμε ότι οι πολίτες, οι πελάτες, μάλλον και ε, οι άλλοι που επωφελούνται από τα στοιχεία μας, να μας έχουν εμπιστοσύνη, να ξέρουν ότι κάνουμε δουλειά για εκείνους Και μόνο έτσι σε εμπιστεύεται ο άλλος. Όταν σου δίνει χρήματα για συγκεκριμένη δράση και συγκεκριμένο σκοπό, χωρίς να πλατιάζουμε. 2.600 υπαλλήλου έχουμε ε, και 300 με 400 ε, χρηματοδοτούνται από εναλλακτικέ ανταγωνιστικές πηγές χρηματοδότησης. Όχι από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. στα μοντέλα, στα πρότυπα αυτό ε, που πρέπει να προσέχουμε είναι οι παράμετροι και τα στοιχεία που τους δίνουμε, γιατί το μοντέλο σου βγάζει ότι του δίνεις ως στοιχεία. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να προσέχουμε ποιες είναι οι καλύτερες περιπτώσεις, ποια είναι τα καλύτερα σενάρια και χρειάζεται μελέτη με αυτούς που φτιάχνουν τα μοντέλα και τα πρότυπα, γιατί το ίδιο μοντέλο μπορεί να σου δώσει τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα ανάλογα με τι στοιχεία θα του βάλεις. Αν δείτε άλλωστε και τις διάφορες ενεργειακές ε, προοπτικές, να δούμε ποιοι είναι οι περιορισμοί, ε, τι θέλουν να περάσουν ορισμένες ομάδες συμφερόντων, τι μήνυμα θέλει ο καθένας να σου περάσει. Και πάντα αυτό χρειάζεται ανάλυση και ένα μοντέλο για να βγάλεις ένα καλό σενάριο. Προσπάθησα να καλύψω τις περισσότερες από τις ερωτήσεις σας και σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γενικά, Γενική Διευθυντά, να σας ευχαριστήσω και εξ ονόματος όλων των συναδέλφων μου. Ο συνάδελφος Μπούτικοφ έχει άλλη μια ερώτηση. Ναι, Πρόεδρε, θα μπορούσαμε να μας δώσετε, αν θέλετε, τις ε, διαφάνειες. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Θα σας δώσουμε τις διαφάνειες. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και γι' αυτό, κύριε Διευθυντά. Και σας ευχαριστούμε και για τη συζήτηση. Και σίγουρα θα επανέλθουμε σε διάλογο και εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και όπως είπε και ο κύριος Τσίτσεστερ, συνέστησε στους συναδέλφους καινούργιου και μη να έρθουν να επισκεφτούν τα κέντρα σας. Και το ξέρω ότι είμαστε ευπρόσδεκτοι πάντα σε εσά. Είναι πολύ σημαντικό το κέντρο και σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε εδώ πέρα σήμερα. Meine lieben äh, έχουμε το θέμα της κινητικότητας ε, των ερευνητών, το οποίο το έχουμε συζητήσει σε πολλές ε, περιστάσεις και πριν από κάποιο καιρό η Επιτροπή ε, ανέθεσε μία έρευνα μία μελέτη για το θέμα της κινητικότητας της διασυνοριακής των ερευνητών. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η μελέτη αυτή και την λάβατε όλοι σας, την έχετε μπροστά σας ε, σε πολύχρωμες διαφάνειες. Θα θέλαμε όμως να γίνει και μια επίσημη παρουσίαση στην ε, Επιτροπή για να ακούσουμε και ποια ήταν τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής. Να καλωσορίσω λοιπόν τον κύριο Μπιλιάμ. Ελπίζω, ελπίζω να τον πρόφερα σωστά το όνομα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν θα μας παρουσιάσετε την μελέτη και μετά θα έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε και κάποιες ερωτήσεις. Θα ήθελα να επικεντρωθούμε, να είναι μάλλον αρκετά συνοπτική η παρουσίαση για να έχουμε και χρόνο να κάνουμε ερωτήσεις μετά. Έχετε το λόγο. Okay. Good afternoon, everybody. Μάλιστα, ευχαριστώ και καλησπέρα σε όλους. Κίμω Βιλιάμα ονομάζομαι και είμαι εκπρόσωπος ε, τον ε, υπεύθυνο για τη μελέτη αυτή. Τα άλλα τα ονόματα τα βλέπετε στη διαφάνεια. Θα ήθελα καταρχάς να μιλήσω για το περιεχόμενο της ε, έρευνας και της παρουσίασης. Τα θέματα λοιπόν που πρέπει να καλύψω σήμερα καταρχάς αφορούν την, τα θέματα κινητικότητας των ε, ρευνητών, των νέων και κάποιες συστάσεις για το πώς μπορεί να διευκολυνθεί η κινητικότητα των νεαρών ερευνητών στο μέλλον. Καταρχάς να αναφέρω κάποια βασικά κάποια βασικά στοιχεία. Τι εννοείται με την κινητικότητα ερευνητών κατά δεύτερον. Γιατί είναι σημαντική η κινητικότητα των ερευνητών. Θα κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις για την κατάσταση στην κινητικότητα των ερευνητών στην Ευρώπη σήμερα. Θα αναφερθώ στις βασικές προκλήσεις Θα εξετάσω επίσης εν συντομία κάποια μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιες πρωτοβουλίες. Θα δώσω κάποια παραδείγματα. Ένα παράδειγμα που ονομάζεται ε, χάρτης και κώδικας και στο τέλος θα καταλήξουμε σε κάποιες σύντομες συστάσεις. Να ξεκινήσω λοιπόν αναπτύσσοντας το τι είναι η κινητικότητα των ερευνητών. Γενικά, είναι διαφορετική κινητικότητα από τη μετανάστευση. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Κάπου αναφέρεται ότι μιλάμε για την ελεύθερη μετακίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι για την μετανάστευση Δηλαδή, η κινητικότητα περιλαμβάνει και κάποια κυκλοφορία, μια κίνηση ατόμων. Όχι απλά τη μετανάστευση σε μια άλλη χώρα μόνιμα. Επίσης, έχουμε την μακροπρόθεσμη και ε, βράχυπρόθεσμη κινητικότητα. Βράχυπρόθεσμη κινητικότητα κάποιες εβδομάδες εννοείται, κάποιες ημέρες, κάποιους μήνες, ενώ η μακροπρόθεσμη κινητικότητα είναι από ένα έως και περισσότερα χρόνια. και στη συνέχεια πρέπει να διευκρινίσουμε ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές ως προς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στα δύο είδη κινητικότητας. Ε, στη συνέχεια είναι σημαντικό να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ της ε, κινητικότητας έξωθεν, δηλαδή το, την έλξη ερευνητών από το εξωτερικό και την ε, κινητικότητα προς τα έξω, δηλαδή τους ερευνητέ οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό. Και αυτό ισχύει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή ένωση Εξετάζουμε δηλαδή πόσοι έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι προβλήματα έχουν τα άτομα που έρχονται από τρίτες χώρες και φυσικά πού κατευθύνονται οι ερευνητές που φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που είναι σημαντικό επίσης είναι να διαχωρίσουμε τα θέματα σωματικής κινητικότητας, πραγματικής κινητικότητας και της εικονικής κινητικότητας. Γιατί η πραγματική κινητικότητα είναι και χρονοβόρα και κοστίζει χρήματα. Ενώ οι δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία πληροφορίας είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες σε ό,τι αφορά την εικονική κινητικότητα. Φυσικά δεν αντικαθιστά αυτό την πραγματική κινητικότητα, αλλά την συμπληρώνει. Και τέλος, έχουμε την διατομεακή κινητικότητα, δηλαδή μεταξύ ακαδημαϊκού κόσμου και βιομηχανίας και μεταξύ διαφορετικών τομέων, διαφορετικών ε, ειδικεύσεων στους ακαδημαϊκούς κύκλους. Σήμερα κυρίως μιλάμε για την ε, διαπεριφερειακή διασυνοριακή σωματική, πραγματική δηλαδή κινητικότητα των ε, ερευνητών νεαρής ηλικίας. Γιατί λοιπόν είναι σημαντική η κινητικότητα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές οικονομικές μελέτες για την ακριβή προστιθέμενη αξία της κινητικότητας. για να υπάρχουν δηλαδή και στατιστικά στοιχεία. Αλλά έχουν εντοπιστεί στις ε, μελέτες πολλά θετικά στοιχεία κατά το παρελθόν, καταρχάς κοιτώντας την αγορά εργασίας. Θα μπορούσε... Μάλλον η κινητικότητα θα μπορούσε να δώσει μια καλύτερη αναλογία μεταξύ ε, προσφοράς και ζήτησης ερευνητών στην Ευρώπη και αυτό είναι σημαντικό γιατί διάφορες χώρες, οι διάφορες περιφέρειες έχουν συγκεκριμένες ανάγκες για συγκεκριμένους ε, ε, ειδικού και σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν αυτοί οι ειδικοί στην περιφέρεια όπου χρειάζονται. Έτσι λοιπόν με την κινητικότητα ε, υπάρχει μεγαλύτερη εξειδίκευση και βελτίωση της απόδοσης της έρευνας. Της έρευνας. Επίσης θα είναι πιο ανοιχτή η... Μάλλον, αν είναι πιο ανοιχτή η αγορά για την κινητικότητα των ερευνητών, αυτό σημαίνει ότι έχουμε πιο πολλές δυνατότητες για την ίδρυση κέντρων αριστείας. στην Ευρώπη. Άρα η συσσόρευση κρίσιμης μάζας είναι σίγουρα μία από τις, ε, ένα από τα πλεονεκτήματα της κινητικότητας. Ο κόσμος δηλαδή να μπορεί να δουλέψει εκεί όπου χρειάζεται η ειδικότητά του. Επίσης, ε, ένα άλλο πλεονέκτημα, η καλύτερη αντιστοίχηση θέσεων εργασίας για το εργατικό δυναμικό Υψηλή εξειδίκευση, γιατί το εργατικό δυναμικό αυτό δεν ε, βρίσκει απαραίτητα θέση εργασίας στη χώρα του. Με την κινητικότητα λοιπόν δίνεται η δυνατότητα να ακολουθήσει κανείς μια πιο λαμπρή καριέρα ως ερευνητή. Επίσης, ε, η καλύτερη έρευνα στα πλαίσια της συνεργασίας και μεταφορά γνώσης. Αυτό που αναφέρετε και εσείς προηγουμένως. Η γνώση μπορεί να ρέει πιο εύκολα μεταξύ των διαφόρων α, ομάδων έρευνας. Και επίσης η, τα καινούργια στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα μπορούν να εφαρμόζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο γρήγορα. από ευρύ, υπό ευρύτερο πλαίσιο τώρα, από πλευρά τη ανταγωνιστικότητα, ε, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για άτομα υψηλή εξειδίκευση. Γιατί η οικονομία της γνώσης απαιτεί πιο εξειδικευμένους ερευνητέ. προκειμένου να είναι ανταγωνιστική η οικονομία. Και αυτό αφορά και τη γύρανση του πληθυσμού, που επίσης ε, επηρεάζει τους ερευνητές. Γιατί όταν υπάρχει γύρανση και στους ερευνητέ, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ζήτηση και ανάγκη για νεαρότερους ερευνητέ. Και επίσης ένας άλλος σχετικός παράγοντας είναι ο λένε και αυξανόμενος παγκόσμιος ανταγωνισμός για τα ταλέντα, για τα μεγάλα μυαλά. Και ως τώρα η Ευρώπη δεν έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία στον διεθνή αυτό ανταγωνισμό. Τώρα, δεν έχουμε αριθμητικά στοιχεία, αλλά βλέπετε στη διαφάνεια ότι υπάρχει κάποια κατάταξη. Έχουμε κάνει κάποια κατάταξη των χωρών βάσει πρόσφατης μελέτης. Μιας μελέτης που έγινε για το IPTS που είναι μέλο, μέρος του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Και όπως βλέπετε είναι πολλές οι χώρες όπου υπάρχει, όπου είναι μάλλον χαμηλή η κινητικότητα η έξωθεν. Αυτό τι σημαίνει ότι δεν είναι τόσο ενδιαφέρουσες οι χώρες αυτές ως πόλος έλξης για τους ερευνητές. Μεγάλη η ομάδα αυτή. Μπορεί κάποιες χώρες να λείπουν από τον κατάλογο, αλλά λίγο πολύ αυτές είναι. Κάποιες άλλες χώρες ε, έχουν σημαντική κινητικότητα προς τα έξω, δηλαδή brain drain, διαρροή εγκεφάλων. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για μικρές χώρες με μικρές γλώσσες όπου είναι ίσως δύσκολο να προσελκύσουν μεγάλες ομάδες ερευνητών. Οπότε φεύγουν πάρα πολλοί ερευνητές από, χώρες, από τις χώρες αυτές και πάλι έτσι υπάρχει ροή της γνώσης και αναπτύσσονται δίκτυα. Το θετικό είναι το εξής. Η κινητικότητα αυξάνεται σε πάρα πολλές ε, χώρες σε αντίθεση με κάποιες άλλες όπου μειώνεται. Και παρά τη γενική αυτή τάση αύξησης ε, της κινητικότητας, οι μελέτες, οι πρόσφατες καταδεικνύουν ότι υπάρχουν ακόμα πολλά εμπόδια. Και βλέπετε λοιπόν κάποιες από τις βασικές προκλήσεις, κάποια από τα βασικά προβλήματα. Καταρχάς σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση της κινητικότητας και τους μισθούς. Πρόκειται για το πιο σημαντικό πρόβλημα. Και κυρίως μιλάμε για συγκριτικό πρόβλημα σε σχέση με την ε, τρέχουσα αμοιβή των ερευνητών αυτών. Η κινητικότητα με βραχυπρόθεσμα συμβόλαια δεν είναι πάντα ανταγωνιστική. Και η χρηματοδότηση έχει να κάνει συχνά με το ίδρυμα που προσλαμβάνει τους ερευνητές. Και επίσης έχει να κάνει και με το έμεσο κόστος της κινητικότητας. Και όλα αυτά καθιστούν την κινητικότητα κατά το πιο ε, επικίνδυνο, ιδιαίτερα για τους νέους. Κάτι άλλο, το οποίο συζητάμε τα τελευταία χρόνια είναι τα θέματα κοινωνικής ασφάλειας και τα θέματα συνταξιοδότησης. Η δυνατότητα δηλαδή να διατηρηθούν αυτά τα δικαιώματα και να μεταφερθούν τα δικαιώματα αυτά. Ιδιαίτερα για ερευνητέ που επιδεικνύουν υψηλή κινητικότητα. Αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια για την ε, μετακίνηση αυτή των ε, ερευνητών. Έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα, αλλά αυτό εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πρόβλημα. Στη συνέχεια, ιδιαίτερα για τους νέους ισχύει αυτό, η έλλειψη δυνατοτήτων για ανάπτυξη της καριέρας τους. Θεωρείται ένα από τα βασικά προβλήματα. Σε πολλές χώρες φαίνεται ότι, υπάρχουν, ότι θέματα αρχαιότητας, τα οποία ουσιαστικά είναι απαγορευτικά για νέους ανθρώπους να έρθουν και να εγκατασταθούν δηλαδή στα ευρήματα αυτά. Επίσης τα θέματα τα γλωσσικά. Από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τη μελέτη δεν αποτελεί αυτό βασικό πρόβλημα γιατί είναι ούτως ή άλλως διεθνές το περιβάλλον και πολλά γράφονται σε μια βασική γλώσσα. Πιο πολύ υπάρχουν προβλήματα κοινωνικής ζωής αν θέλετε κοινωνικού περιβάλλοντος και σε κάποιες περιπτώσεις ε, το θέμα της γλώσσας είναι λίγο πιο σημαντικό από ότι σε άλλες. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Τώρα, η μη αναγνώριση της εμπειρίας της κινητικότητας κατά την ανάπτυξη της καριέρας. Αυτό για τους νέους είναι μεγάλο πρόβλημα. Πάντα είναι, ενέχει κάποιους κινδύνους η μετακίνηση, η κινητικότητα. Το να επιλέξει κανείς να μην μείνει στην πατρίδα του και να συνεργαστεί με τους καθηγητές του εμπεριέχει κινδύνους. Το να φύγει, να πάει στο εξωτερικό, να χάσει τις επαφές του. Ιδιαίτερα αν δεν θεωρείται αυτό ως κάτι στο βιογραφικό σημείωμα. Επίσης, η έλλειψη πληροφόρησης. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δημιουργηθούν διάφορες υπηρεσίες ε, πληροφόρησης, αλλά παρόλα αυτά οι θέσεις που ανοίγουν σε άλλες χώρες δεν ε, τις γνωρίζουν απαραίτητα όλοι. Δεν γνωρίζει δηλαδή ο καθένας τι δυνατότητες έχει σε κάθε χώρα. Επίσης, η έλλειψη ανοιχτού και ανταγωνιστικού συστήματος προσλήψεων σε διεθνές επίπεδο. Σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές χώρες, οι διαδικασίες δεν είναι διαφανείς και ανοιχτές. Δεν ε, διατίθεται η σχετική πληροφόρηση και ενημέρωση διεθνώς. Οι, επίσης, οι κανόνες μετανάστευσης έχουν σημειωθεί κάποια βήματα προόδου ως προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά πολλοί νεαροί θεωρούν ότι αυτό αποτελεί σημαντικό πρόβλημα ακόμη, ιδιαίτερα αν προέρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κάποια θέματα ε, συμβατικά και νομικά. Θέματα, για παράδειγμα, μεταφοράς ε, χρηματοδότησης και πόρων, τα βράχη πρόθεσμα συμβόλαια. Και αυτά αποτελούν ένα βασικό πρόβλημα, γιατί είναι οι συμβάσεις αυτές οι βραχυπρόθεσμες το πιο συνηθισμένο φαινόμενο για τους νεαρούς ερευνητές. Τέλος, σε κάποιες χώρες που δεν έχουν τόσο ελκυστικά συστήματα έρευνας, διαπιστώνεται μια προθυμία, γιατί δεν θέλουν οι χώρες αυτές να χάσουν τους ταλαντούχους νέους ερευνητές τους, που ενδεχομένως να φύγουν στο εξωτερικό και να μην ξαναγυρίσουν. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο αποτυπώνει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ε, ερευνητικών δομών, των ερευνητικών ε, πόρων και συστημάτων μεταξύ των διαφορετικών χωρών. Να εξετάσω γρήγορα τώρα κάποια ευρωπαϊκά μέτρα που υπάρχουν. Το πρόγραμμα πλαίσιο, το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο για την έρευνα αυτή. Ευρωπαϊκός Χάρτης για ερευνητέ και χάρτης, ε, συγγνώμη, κώδικας διοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία εθελούσια η οποία καθιερώθηκε το 2005 προκειμένου να καταστεί η πρόσληψη και σχετικέ πρακτικέ για την πρόσληψη πιο δίκαιε για τι διάφορε χώρε. Και η διαδικασία τη Μπολόνια εν μέρη επηρεάζει την κινητικότητα γιατί προβλέπει συμβατότητα μεταξύ των πτυχίων μεταξύ των κρατών μελών. Άρα είναι πιο εύκολη η σύγκριση. Επίσης υπάρχει και μία οδηγία για να εγκριθεί μία θεώρηση επιστημονική για ερευνητές τρίτων χωρών προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες ε, πληροφόρησης οι οποίες ε, ξεκίνησαν με το πρόγραμμα ERAMOR με τον κόμβο κινητικότητα των Ευρωπαίων ερευνητών με το Euraccess το οποίο αφορά τις ΕΠΑ και ενημερώνει για τις δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρόσφατα μια νέα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση μια εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των απαραίτητων ε, ερευνητών και προτείνονται δράσεις σε τέσσερις βασικούς τομείς. Αυτή είναι η πλέον πρόσφατη πρωτοβουλία με σκοπό να επιταχύνει την όλη διαδικασία η οποία ήδη έχει ξεκινήσει κατά το παρελθόν. Ένα παράδειγμα για τις πρόσφατες αυτές ε, πρωτοβουλίες. Είναι καλό παράδειγμα για όλα τα προβλήματα που αφορούν την κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ονομάζεται Charter and Code, χάρτης και κώδικας. Κοιτώντας τις διάφορες ε, οργανώσεις που έχουν ε, υιοθετήσει αυτό το Charter and Code στην Ευρώπη. Φαίνεται ότι λίγες είναι οι οργανώσεις που έχουν υπογράψει ή έχουν εγκρίνει τον χάρτη αυτό σε διάφορες χώρες και αυτό καταδεικνύει ότι στηριζόμαστε κυρίως στις εθελοντικές δράσεις των ε, κρατών μελών και παρόλο που υπάρχει πρόοδος, είναι πάρα πολύ αργή αυτή η πρόοδος, το οποίο μας οδηγεί στη φάση των συστάσεων. Φαίνεται ότι τα μέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, από μόνα τους δεν αρκούν για να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια για την κινητικότητα των ερευνητών. Υπάρχουν πολλές καλές ε, ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες οι οποίε ξεκίνησαν την τελευταία δεκαετία. Το πρόβλημα είναι ότι χωρί τα κράτη-μέλη, χωρί την ενεργό συμμετοχή τους στις δραστηριότητες αυτές, αν αυτές οι νέε πρωτοβουλίε δεν εφαρμοστούν από τα κράτη-μέλη, η όλη διαδικασία, η όλη πρόοδος θα είναι πάρα πολύ άνηση και πολύ αργή. Και βλέπουμε ότι σε κάποιες χώρες εφαρμόζονται αυτές οι νέες καινούργιε πρωτοβουλίε και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι σε άλλε χώρε. Για να διασφαλίσουμε λοιπόν την ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών, χρειαζόμαστε μια εταιρική σχέση με τους ερευνητέ. Αυτό αποτελεί ένα από τα σημεία κλειδί. Κάτι άλλο. Να αντιμετωπιστούν θέματα κοινωνικής ασφάλειας και συνταξιοδότησης. Υπάρχει νομοθεσία η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει την μεταφορά του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης για τους ερευνητέ. Το πρόβλημα είναι μάλλον η διοικητική συνεργασία μεταξύ των χωρών. Οι οργανώσεις ερευνητών και οι ίδιοι ερευνητέ γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν. Είναι θέμα ενημέρωσης. Η έγκριση τώρα του Charter and Code προκειμένου να καταστεί η αγορά πιο διαφανής και πιο ανταγωνιστική σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Όλα αυτά θα πρέπει να προχωρήσουν περαιτέρω προκειμένου όχι μόνο να προσυπογράψουν με οργανώσεις αλλά και να εφαρμόσουν το χάρτη αυτό στην πράξη στη συνέχεια θα πρέπει να ξεπεραστούν τα οικονομικά προβλήματα, τα οποία πλήττουν κυρίως τους ε, νέους ερευνητές. Προκειμένου, για παράδειγμα, να μπορεί να μεταφέρει κανείς την επιδότησή του. Η υποστήριξη, η να μην αποτελεί πρόβλημα για τα ιδρύματα υποδοχής και κάποιοι ανέφεραν κάποια βάουτσερ για την κινητικότητα των ερευνητών το οποίο τι σημαίνει πέρα από την χρηματοδότηση, πέρα από το μισθό, να υπάρχει και χρηματοδότηση όλων των έμεσων εξόδων. Για παράδειγμα, για τη φύλαξη των παιδιών, για την ε, έβρεση κατοικίας, όλα αυτά τα θέματα που μπορεί να πλήττουν τους ε, νέους ερευνητές, ιδιαίτερα όσους έχουν οικογένεια. Στη συνέχεια, μέτρα για την αύξηση της κινητικότητας ερευνητών από τρίτες χώρες. θα πρέπει τα κράτη-μέλη να παρατρινθούν να εφαρμόσουν το πακέτο επιστημονικής θεώρησης και επιδοτήσεις ε, για την, να δοθούν επίσης επιδοτήσεις για την επιστροφή ε, ερευνητών, γιατί υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλοί ερευνητές οι οποίοι έχουν μείνει στη ΣΥΠΑ. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος. Στη συνέχεια, ενσωμάτωση και κινητικότητα ερευνητών με άλλα μέτρα υποστήριξης της καινοτομίας. Υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα και φυσικά η κινητικότητα δεν πρέπει να θεωρηθεί μεμονωμένη. Πάντα ε, διασυνδέεται με άλλες πρωτοβουλίες. Και επίσης αυτό που σε πολλές περιπτώσεις έχει σημειωθεί ότι λείπουν αξιόπιστα στοιχεία, μια αξιόπιστη βάση δεδομένων προκειμένου να καταμετρηθεί και ο αντίκτυπος της κινητικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι δύσκολο να καταγράψουμε την εξέλιξη της κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση. Ο συνάδελφος Τσουκαλάς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη προσοχή άκουσα την έκθεση για την κινητικότητα των ερευνητών είναι κρίμα που οι συνάδελφοι απουσιάζουν σήμερα, επειδή η προηγούμενη παρουσίαση του Γενικού Διευθυντή του GRC, συνδυασμένη με την έκθεση για την κινητικότητα που μόλις τώρα ακούσαμε, συνδυασμένη με τα όσα ακούστηκαν επί δύο ημέρες στο First European Innovation Summit, συνδυασμένη με τη διακήρυξη του Λούντ και τα trends το 2025, συνδυασμένη με την αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας, συνδυασμένη με την πραγματική επικράτηση στην έρευνα των χωρών που δεν είναι στην Ευρώπη, κάνει αυτή τη συζήτηση πολύ επίκαιρη. Η μελέτη που μόλις μας γνωστοποιήθηκε φύγει με μεγάλη επάρκεια τις αιτίε για τις οποίες ε, υπάρχει μειωμένη κινητικότητα στο ευρωπαϊκό επιστημονικό δυναμικό. Αυτό που δεν γνωρίζω είναι αν αυτά τα μέτρα που στο τέλος παρουσιάζονται ως conclusions ή recommendations όπως είδα τώρα, θα μπορούσαν να έχουν μια πολύ πιο πρακτική και αποτελεσματική μορφή. Η τη λέει σε ένα σημείο ότι θα έπρεπε να πιεστούν περισσότερο οι κατηδίαν χώρα τα μέλη κράτη, ώστε να εφαρμόσουν τον... Αυτό ίσως θα μπορούσε να ε, γίνει με συγκεκριμένη λήψη μέτρων, δεν ξέρω ποιος μπορεί να τα πάρει. Όμως η Επιτροπή μας, η οποία είναι υπεύθυνη για την έρευνα, νομίζω ότι έχοντας όλα αυτά υπόψη, πρέπει να κάνει κάτι πιο ε, ε, πιεστικό προς τα κατάλληλα τα αρμόδια κοινοτικά όργανα, ώστε το ζήτημα της έρευνας να μην αποτελεί πια ένα ιδεολόγημα το οποίο επαφίεται σε μελέτες ή στρατηγήματα. Οι αριθμοί είναι πολύ σαφείς το 60% του επιστημονικού, συνολικού επιστημονικού αποτελέσματος παράγεται στην Αμερική. 62% του γραπτού επιστημονικού λόγου είναι στην αγγλική γλώσσα και το 80% είναι στην Αμερική. 80% των νομπελιστών είναι στα 60 πανεπιστήμια της Αμερικής, τα οποία παράγουν το 60% της του αμερικανικού επιστημονικού outcome, δηλαδή το 36% του παγκόσμιου. 25% περίπου, αν θυμάμαι καλά, είναι οι διεθνείς πατέντες που έχει η Αμερική και συνεπώς, εάν θέλουμε κάτι να κάνουμε, θα πρέπει να το κάνουμε πιο ριζοσπαστικά. Είναι προφανές ότι μας λείπει κάτι. Ε, και μας λείπει κάτι, όχι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάνει πολλά. Έχει κάνει πολλά, έχει ενοποιήσει το ζήτημα το, ξέρουμε πια ποιο είναι το πρόβλημα, αλλά μας χρειάζεται κάτι ακόμα. Ίσως η Επιτροπή μας θα έπρεπε κάτι να κάνει προς αυτή την κατεύθυνση. Γνωρίζουμε ότι είναι πια μεγάλη ανάγκη να επενδύουμε στην αριστεία. Ξέρουμε ότι ποσοτικά δεν φτάνει το να δίνουμε χρήματα. Ξέρουμε ότι σήμερα οι όροι παραγωγής ζητούν όλο ένα καλύτερα προϊόντα, φθηνότερα προϊόντα και αυτό μπορούν να το πράττουν μόνο οι άριστοι. Επομένως, η αριστεία δεν είναι ηθικού τύπου πρόταγμα. Είναι οικονομικού, οικονομικού τύπου ανάγκη. Αυτή την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση την έχει πάρει είδηση, όμως παράγοντες όπως είναι η κινητικότητα εμποδίζουν την ανάπτυξη ενός πλέγματος δράσεων και αποτελεσμάτων που θα έφερναν την Ευρώπη στο σημείο που οραματίστηκε μάλλον επιπόλαια η διακήρυξη της Λισαβόνας που μας ήθελε την πρώτη οικονομία το 2010 βασισμένη σε μια οικονομία της γνώσης. Αυτή η συγκεκριμένη οικονομία της γνώσης που λέμε ότι βασίζεται και καλά το λέμε στο τρίγωνο της γνώσης, δηλαδή education, research και innovation πρέπει να υποστηριχθεί full steam. Δεν γνωρίζω τον τρόπο κύριε Πρόεδρε. Ε, είμαι βέβαιος ότι με μια πιο λεπτομερή συζήτηση αυτή η Επιτροπή θα έπρεπε να καταλήξει σε κάποια μέτρα που θα πρότεινε στο Κοινοβούλιο για το πολύ επίγον ζήτημα και με συγχωρείτε που δεν εσιάστηκα στην πολύ άρτια αυτή καταγραφή της πραγματικότητας αλλά ήταν όλα μαζί μαζεμένα που μου δώσαν το τοπίο. Ευχαριστώ äh, Σας ευχαριστώ και εγώ. Θα μου επιτρέψετε μια ενδιάμεση πρόταση. Έχετε 100% δίκιο. Ίσως θα πρέπει στην Επιτροπή μας να σκεφτόμαστε κιόλας να αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο σε τέτοιες συζητήσεις. Τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ χρόνο βάλαμε στην ενέργεια, στις κλιματικές συζητήσεις. Στο μέλλον ίσως να σκεφτούμε μήπως να αλλάξουμε λίγο το κέντρο βάρους μας στην Επιτροπή. Αυτό απευθύνεται σε όλους τους συναδέλφους και τους συντονιστές για το πώς θα ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Παρακαλώ και τη Γραμματεία να το σημειώσει αυτό που είπατε και να το ξανακοιτάξει. Οπωσδήποτε του χρόνου να είναι προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ ειλικρινά. Έχω ζητήσει και άλλη το λόγο. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Κυρία Γκουτιέρες Κορτίνες, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Πρώτον, μπαίνω στο ψητό. Ευχαριστώ που ήρθατε. Εκπλήσωμαι που δεν βάλετε κάποιες αξίες που βάλαμε εμείς και στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και σε προηγούμενα σε συστάσεις και έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράδειγμα. Με έμεσο τρόπο μπορεί να το λέτε, αλλά επειδή δεν θέλουν να τα ακούσουν οι χώρες, γιατί το πρόβλημα είναι των κρατών φυσικά, δεν τους αρέσει. Δεν ξέρω, ίσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θεώρησε ότι ήταν ε, αρκετό το Marie γιατί χαίρονται όλοι και είναι κατεθουσιασμένοι, αλλά δεν είναι καθόλου επαρκές, είναι πολύ χαμηλό το ποσό. Λοιπόν, δεν υπάρχει σαφής αναγνώριση εδώ της αξίας της έρευνας στις χώρες μας. Στη σταδιοδρομία για τον ερευνητή και το πώς αξιολογούνται πώς δίνονται οι θέσεις, οι ερευνητικές. Δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο. Είναι πολύ καλύτερο να είναι κανείς εκτός της Ένωσης παρά εντός. Θα πρέπει να βάλουμε κριτήρια. Γιατί ξέρω ανθρώπους που έχουν πάει 15 μέρες διακοπές στο Εδιμβούργο με τη γυναίκα τους, πέρασαν και από το πανεπιστήμιο, πήραν ένα χαρτάκι και νομίζουν ότι είναι εντάξει. Και όλος έχει κάνει σπουδέ ολόκληρε. Ε, ε, θα πρέπει, καλή είναι η κινητικότητα, αλλά θα πρέπει να έχουμε κριτήρια. Υπάρχει ένα κίνδυνος ενδογαμίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει μελέτες στα κράτη-μέλη τι γίνεται. Για παράδειγμα, στι Ηνωμένε Πολιτείε ή στο Ισραήλ, το διδακτορικό σου, όταν το κάνει ένα πανεπιστήμιο, απαγορεύεται να δουλέψει στο ίδιο πανεπιστήμιο. Στι λατινογενεί χώρε τη Λατινική Αμερική είναι το αντίστροφο. Όποιο δεν κάνει διδακτορικό στο πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να μπει με τίποτα στη συνέχεια ως ερευνητή, διότι υπάρχει ο καθηγητής τη Έδρα και τον έχει σαν παιδί του μετά τον φοιτητή του διδακτορικού και ε, υπό την προστασία του, την επίβλεψή του και ακολουθεί καριέρα. Επίσης υπάρχουν ε, και ψευδή βιογραφικά. Πλαστογραφούνται πολλές φορές τα βιογραφικά στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν ερευνητικέ ομάδε ανύπαρκτες που φαίνονται στα χαρτιά και κάποιο κάνει μαθήματα και εμφανίζεται ότι είναι ερευνητή. Εντάξει, και αυτό να το σκεφτούμε. Λοιπόν, πριν από 15 χρόνια λέγαμε στα πανεπιστήμια την αξιολόγηση, την αμοιβαία βαθμολόγηση και έγινε πόλεμος αμήλικτος έτσι ώστε τα καημένα τα παιδιά που πηγαίναν στον έρασμο, οι φοιτητέ να μπορέσουν να του αναγνωρίσουν τον τίτλο και το πτυχίο του στα πανεπιστήμια. Αδυσόπιτος πόλεμος έγινε για να περάσει αυτό από τα πανεπιστήμια. Λοιπόν, μπορεί κάποιο να έχει πάει σε ένα πανεπιστήμιο, να έχει κάνει ένα μάστερ, ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό. Και τα ποιοτικά ε, μάστερ θα πρέπει να τα ελέγχει η Ευρώπη. Να ζητάμε από τις κράτες μέλη να ανοίξουν τα παράθυρα ανοιχτά. Δεν είναι κλειστά αυτά τα ιδρύματα σαν μοναστήρια ε, γυναικεία που απαγορεύεται να πατήσει άνδρα στο πόδι του. Να ανοίξουν τα πανεπιστήμια, να ανοίξουν τις διαδικασίες τους, να αξιολογούνται, να ελέγχονται για να μην ευρεωθεί η μετριοκρατία που υπάρχει σε πολλά μέρη. Και το χειρότερο πράγμα που μπορεί κανείς να έχει στη ζωή του είναι να, περιστοιχίζεται από μετρίους. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτά που λέω. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος για το σθένος ε, και το πάθος σας. Η κυρία Ρία Χωρίς μικρόφωνο, δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την παρουσίαση του. Είναι γεγονός και συμφωνώ με τον Πρόεδρο. Επανειλημμένα έχουμε συζητήσει για την κινητικότητα εδώ, αλλά είναι από τα βασικά θέματα που πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας αν θέλουμε να δώσουμε μια σημαντική όθηση στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και συμφωνώ με τον Πρόεδρο. Θα πρέπει να ασχολούμαστε πιο συχνά με τα θέματα αυτά και πολύ επίκαιρη είναι όντω η έκθεση. Μιλήσατε για την κινητικότητα των ερευνητών. Ε, δύο είναι για μένα τα βασικότερα θέματα. Πρώτον, επιγόντως θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ενιαία αγορά ερευνητών και ερευνητριών για ένα μοναδικό ενιαίο μοντέλο σταδιοδρομία στην έρευνα στην Ευρώπη. Και στη συνέχεια θα ήθελα επίσης να τονίσω την ανάγκη να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης για ε, τις συμβάσεις, για την προσφορά, για την προκήρυξη θέσεων ερευνητών παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ωραία το εξηγείτε στην έκθεσή σας και συμφωνώ απολύτως ότι δεν είναι καθόλου εύκολο κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ ε, αργή, χρονοβόρα, πολύ περισσότερο από όσο θα επιθυμούσαμε. Συμφωνώ όμως με ένα από τους προλαλήσαντες, δεν έχουμε πρακτικές ιδέες για να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν θα επαναλάβω τα όσα είπαν οι συνάδελφοί μου, τα ε, συμμερίζομαι. Μερικές ερωτήσεις πολύ συγκεκριμένες τώρα για τα συμπεράσματα. Καταρχάς, μας λέτε ότι τα θέματα του φίλου φαίνονται ως ίσονος σημασίας. Από ό,τι θεωρούσε κανείς αρχικά, μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό γιατί δεν το κατάλαβα. Και ένα δεύτερο ζήτημα, πάλι στα συμπεράσματα, από τη μια λέτε ότι για να διευκολυνθεί η κινητικότητα χρειάζεται αλλαγή στην οτροπία. Να αφήσουμε στην άκρη αυτό που λέτε εθνικές προκαταλήψεις. Και θα πρέπει να είναι η κινητήρια δύναμη η έρευνα, το αντικείμενο της και η κοινή σταδιοδρομία. Μέχρι εδώ συμφωνούμε. Από την άλλη όμως λέτε ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν εργαλεία και μέσα και το εξήγησατε και προφορικά που να διευκολύνουν την επιστροφή στη χώρα προέλευσης των ερευνητών για να αποφευθεί η διαρροή εγκεφάλων, brain drain. Μα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αφού θέλουμε να έχουμε ε, αλλαγή νοοτροπίας και να οικοδομήσουμε ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό χώρο, είναι ενίος ο χώρος. Καλύτερα να αλλάξει η νοοτροπία, να έχουμε κοινή ε, σταδιοδρομία με προοπτικές και το θέμα δεν είναι αν επιστρέφει ο καθένας στη χώρα του στον ενίο ερευνητικό χώρο και από χρηματοδότηση πώς τα βλέπετε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκίρεκ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όταν μιλάμε για κινητικότητα πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε αυτήν που στηρίζεται στην επιστήμη και στην φυγή των, κεφαλ... Ε, ε, εγκεφάλων, brain drain. Είναι όπως την κατάσταση εργοστασίων, το brain drain. Διότι αν εσωτερικά μέσα στην Ένωση ενώ βλέπουμε πάρα πολύ brain drain αυτό δεν είναι θετικό αυτό ε, μειώνει την ισχύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ερευνητικών κέντρων Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να τραβήξουμε μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ της υγιούς κινητικότητας και της φυγής εγκεφάλων, brain drain, όταν οι πραγματικοί επιστήμονες αποφασίσουν να μετακινηθούν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αυτή για κινητικότητα, αλλά πρέπει να έχουν ένα στόχο, έναν επιστημονικό στόχο, όχι μόνο οικονομικό στόχο, όχι να αποφασίσουν να φύγουν μόνο για κάποιους οικονομικούς λόγους. Επιστημονικό στόχος λοιπόν επιβάλλεται, θέλουν να αναπτυχθούν επιστημονικά. Αν όλα τα ακαδημαϊκά κέντρα, τα επιστημονικά κέντρα ήταν στο ίδιο επίπεδο, τότε η κινητικότητα δεν θα είχε νόημα. Γιατί όταν αποφασίζει κάποιο να μετακινηθεί, να μεταφέρει την επαγγελματική του έδρα, α πούμε, ψάχνει το άτομο να βρει ένα μέρος όπου θα αναπτυχθεί καλύτερο, θα έχει καλύτερες συνθήκες για τη δουλειά που του αρέσει να κάνει. Έχουμε λοιπόν, αν έχουμε καλά εξειδικευμένα κέντρα με σωστή υποδομή, μόνο τότε με τέτοια κέντρα θα έχουμε και αξιοπρεπή επαρκή κινητικότητα. Η κινητικότητα για την κινητικότητα είναι άχρηστη. Γιατί ξέρουμε ότι σήμερα δεν χρειάζεται πολύ να μετακινηθεί πολίτη. Έχουμε ένα σωρό ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνία σήμερα. Κατ' εμέ λοιπόν η κινητικότητα για την κινητικότητα θα πρέπει να συνοδεύεται από μια πολλές φορές ακριβή εξειδίκευση στα ανεξάρτητα επιστημονικά κέντρα. Μόνο τότε θα έχουμε μίζωνα ωφέλη από την επιστημονική κοινότητα στο σύνολό της. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ματίας, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον ομιλητή μας για την παρουσίασή του και για όλα τα νούμερα που μας έδωσε και τα δεδομένα. Δεν θα ήθελα να επανελάβω αυτό που είπαν και οι συνάδελφοι. Όλα αυτά ήταν ενδιαφέροντα. Θέλω όμως να δούμε λίγο τις διαφορές που υπάρχουν από χώρα σε χώρα όσον αφορά την κινητικότητα. Αυτές οι διαφορές αντικατοπτρίζουν τις διαφορές που υπάρχουν στο επίπεδο των επενδύσεων στο ΑΕΠ, σε ποσοστό του ΑΕΠ στην κάθε χώρα, Παρά τις συμφωνίες και τις καλές προθέσεις, αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν πολλές διαφορές στα, στις συνθήκες εργασίας, στα συμβόλαια εργασίας. Πολλές φορές η κατάσταση είναι επισφαλής για τον εργαζόμενο. Κάθε φορά που μιλάμε για κινητικότητα πρέπει να βλέπουμε τις λεπτομέρειες. Γιατί πρέπει να βλέπουμε τις λεπτομέρειες και, και δεν υποτιμώ καθόλου τη σημασία της κινητικότητας. Ο λόγος λέω λοιπόν είναι ότι υπάρχει κίνδυνος να αυξήσουμε τις διαφορές που υπάρχουν στην Ένωση μιλώντας γι' αυτά. Υπάρχουν έπειτα και ανισότητες σε όλο τον κόσμο. Πολλοί ανάφεραν παραδείγματος τον όρο brain drain. Εμένα αυτό με ενισχύει πολύ. Αυτή η φυγή εγκεφάλων. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη διαφορετικές απαιτήσει στην Ένωση για την είσοδο για άτομα που προέρχονται από τρίτες χώρες και έρχονται ως ερευνητές Υπάρχουν να δουλέψουν και σε άλλους χώρους. Αυτές τις ανισότητες το, το λιγότερο που πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίσουμε να μην γίνουν πιο μεγάλες. Έπειτα, πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο για την έρευνα. Μια πρακτική δομή που θα διευκολύνει την κινητικότητα. Και ένα κομμάτι από αυτό είναι τα εργασιακά συμβόλαια. Όλοι ξέρουμε σε σχέση με τα ερευνητικά κέντρα ότι οι αξίες του κράτους μέλους εντυπώνονται στο κάθε κέντρο, στην κάθε χώρα έρχονται άτομα από άλλες χώρες αλλά ο τρόπος απασχόλησής τους, ο μισθός που παίρνουν κλπ. μπορεί να είναι πολύ διαφορετική. Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Αυτές είναι προκλήσεις που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε πολύ συγκεκριμένα. Να ενισχυθεί βέβαια η έρευνα στην Ένωση, να απορροφηθεί η κινητικότητα, αλλά χρειάζονται και υλικέ συνθήκες συγκεκριμένες για να το πετύχουμε αυτό. Μόνο τότε η Ένωση θα έχει μια σωστή πολιτική που θα συμφωνεί και με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη και θα εφαρμόζεται καλύτερα. Και θα μειωθούν και οι ανισότητες στις συνθήκες εργασίας. Αυτό είναι ο σωστός τρόπος για να προχωρήσουμε. Και ένα τελευταίο σχόλιο. έχει δημιουργηθεί σύγχυση μεταξύ κινητικότητα και μετανάστευση. Πολλέ φορέ συμβαίνει αυτή η σύγχυση. Φυσικά πρόκειται για δύο τελείω διαφορετικέ έννοιε. Βέβαια υπάρχει η διάσταση βραχυπρόθεσμη και η μακροπρόθεσμη. Μερικέ φορέ όμω αυτό χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να έχουμε επισφαλή συμβόλαια στην έρευνα σε πολλές χώρες της Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ και κάποιου ε, μήνε είμαι βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στου μήνε λοιπόν αυτού. σε πολλέ περιπτώσει άκουσα διάφορα για την ε, κοινωνία που βασίζεται στην γνώση και στην Ουγγαρία συχνά συζητιούνται τέτοια θέματα. Μάλιστα τόσο συχνά που καμιά φορά έχω την εντύπωση ότι η όλη συζήτηση, ο όλος όρος δεν έχει πλέον κανένα νόημα. Ακούσαμε λοιπόν την παρουσίαση για την ε, κινητικότητα των νέων ερευνητών και θεωρώ ότι αυτό αποτελεί μια πολύ σημαντική σύμβολη για την κινητικότητα και για την κοινωνία της γνώσης. Πρόκειται για μια πολύ λεπτομερή παρουσίαση, μια πολύ λεπτομερή μελέτη, όπου ανακύπτουν με σαφήνεια τα εμπόδια που προκύπτουν ως προς την ε, κινητικότητα σε ό,τι αφορά την ε, κινητικότητα προς τα έξω για την ε, Ουγγαρία, για την Πολωνία και ούτω καθεξής. Βλέπω ότι οι χώρες αυτές έχουν χαμηλά ποσοστά ως προς την κινητικότητα αυτή. Συχνά δεν τονίζεται αυτό αρκετά και σε πολλές περιπτώσεις αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στηρίζει τα κράτη-μέλη αλλά και τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν πολλά για την κινητικότητα σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια, τις ανώτατες σχολές. Αναμένουμε από, το, από, τα προσωπικό, από το ακαδημαϊκό προσωπικό να ε, αναπτύξει την καριέρα του. Και σε πολλές περιπτώσεις ε, εργάζονται τουλάχιστον ένα εξάμεινο στο εξωτερικό. Στην Ουγγαρία όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό για τους νεαρούς ε, καθηγητές της ανώτατες σχολές και όχι μόνο λόγω της οικονομικής κρίσης γιατί οι σχολές αυτές, τα πανεπιστήμια λαμβάνουν όλο και λιγότερη χρηματοδότηση και κρατικές ενισχύσεις τα τελευταία χρόνια το νεαρό προσωπικό των πανεπιστημίων. Ακόμα και αν έχετε τη δυνατότητα να μεταβεί στο εξωτερικό για ένα εξάμεινο, δεν το κάνει τελικά. Εγώ, για παράδειγμα, θα μπορούσα στα πλαίσια του προγράμματος Tempus να περάσω τρεις μήνες στο εξωτερικό. Τελικά όμως δεν έγινε γιατί μου ασκήθηκε πίεση και δεν ε, αξιοποίησα αυτή την ευκαιρία οι κυβερνήσεις ε, μιλάνε συνεχώς και ακατάπαυστα για την κοινωνία που βασίζεται στη γνώση. Χρειαζόμαστε όμως προς αυτό το σκοπό καλύτερη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Χίπνερ. E, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ για την εξαιρετική αυτή παρουσίαση θίξατε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο θα είναι καθοριστικό για το μέλλον της Ευρώπης. Ε, πώς έχει σήμερα η κατάσταση. Έχουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια, πολύ καλούς και δυναμικούς ερευνητές. Δεν έχουμε όμως δομές που να συγκεντρώνουν όλους αυτούς τους ερευνητές προκειμένου σε παγκόσμιο επίπεδο να επιτελέσουν ένα σημαντικό έργο. Το βραβείο Νόμπελ απονέμεται κάθε χρόνο, αλλά δεν ε, βραβεύονται ε, Αμερικανοί ερευνητές. Είναι ε, ερευνητές από όλο τον υπόλοιπο κόσμο που εργάζονται όμως στην Αμερική και τελικά συνδράμουν στην οικονομική επιτυχία της Αμερικής. Αυτό χρειαζόμαστε και στην Ευρώπη. Μια κατάσταση στην οποία οι ερευνητές με καλύτερους όρου έρευνα δεν θα αναγκάζονται να φεύγουν για τι ΗΠΑ τα πιο οι πιο πολλές ε, ε, ερευνητικέ οργανώσει έχουν πολύ πρακτικά προβλήματα και σημαντικά μάλιστα. Ε, χρηματοδότηση των κτηρίων, για παράδειγμα, και ακόμα ιδιαίτερα μάλλον λόγω τη οικονομική κρίση, φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα που αντιμετωπίζει και η βιομηχανία για την παραγωγή. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε, όπως είπε και ο κύριος Γκέρεκ, πώς μπορούμε να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένους τομείς σε διάφορες χώρες και να επενδύσουμε στους τομείς αυτούς προκειμένου να σημειώσουμε επιτυχία στους συγκεκριμένους αυτούς τομείς. Σας ευχαριστώ και πάλι για την καλή αυτή παρουσίαση, αλλά σας παρακαλώ να σκεφτείτε μήπως θα μας κόπιμο να δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα εξαιρετικό ερευνητικό κέντρο προκειμένου να μην μένει πάντα πίσω η Ευρώπη. Γιατί τι παρατηρούμε, ότι ε, οι μαθητές ακόμα κερδίζουν διάφορα ε, σημαντικά βραβεία και τελικά φεύγουν για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Χάνεται τεράστιο δυναμικό, ιδιαίτερα από τις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Το βλέπουμε αυτό και για τους ε, ερευνητές αλλά και για τις οικογένειές τους. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Μάλιστα. Πάρα πολλές ερωτήσεις λοιπόν για τον κύριο Βιλιάμα. Σας παρακαλώ να τις απαντήσετε αν θέλετε να κάνετε σχόλια. Μάλιστα. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος όμως. Μάλιστα. Ωραία. Θέσατε πολλά ζητήματα. Θα προσπαθήσω να σχολιάσω κάποια εξ αυτών. Ένα από τα βασικά θέματα στην όλη συζήτηση για το brain drain, για τη διαφυγή εγκεφάλων, για τη χρηματοδότηση, που τονίζει το γεγονός ότι η κινητικότητα δεν αποτελεί μεμονωμένο παράγοντα. Είναι κάτι το οποίο ε, σχετίζεται με τις δυνατότητες για σταδιοδρομία των νέων και για το πώς, με το πώς μπορούν να αναπτύξουν ενδιαφέρουσες ε, σταδιοδρομίες και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και αυτό αποτελεί μια βασική διαφορά με τη ΣΥΠΑ. Στη ΣΥΠΑ υπάρχουν καλέ σχέσει για τη σταδιοδρομία. Και αυτό μας οδηγεί σε άλλα ζητήματα, σε ό,τι αφορά τους πόρους, για παράδειγμα, και τις υποδομές ε, της έρευνας, τα συστήματα ε, έρευνας. Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και αυτό είναι θεμελιώδου σημασίας. Κάποιες χώρες δεν μπορούν να προσελκύσουν νέους ερευνητές, όχι λόγω της γλώσσας, όχι λόγω των συστημάτων, αλλά επειδή πολύ απλά δεν μπορούν να τους παρέχουν καλές ευκαιρίες έρευνας. Άρα ένα βασικό θέμα που σχετίζεται με την κινητικότητα είναι η ανάγκη να βελτιώσουμε το σύστημα σε πολλές χώρες προκειμένου να είναι πιο αποδοτικό. Δεν μιλάμε μόνο για την κινητικότητα, μιλάμε και για το σύνολο της έρευνας και του επίπεδου της έρευνας. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλε τι ερωτήσει που θέσατε, ωστόσο σε ό,τι αφορά τις πρακτικές λύσεις. Υπάρχουν αρκετέ λύσεις που έχουν εφαρμοστεί σε διάφορες χώρες. Δεν ε, ανέφερα τέτοια παραδείγματα, αλλά υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα και νομίζω ότι μια πιο λεπτομερής ε, μελέτη θα πρέπει να γίνει για τα παραδείγματα αυτά ή τουλάχιστον για το συντονιστικό ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε καλή θέση για να ασκήσει αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μπορεί να παρακολουθήσει τι γίνεται στις ε, με μονομενες χώρες, να αναπτύξει μια εταιρική σχέση μεταξύ των χωρών, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος. Με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, ε, οι καλές πρακτικές μπορεί να διαδοθούν, αν θέλετε, σε όλες τις χώρες. Χρειάζεται λοιπόν συντονισμός. Συντονισμός κάποιου είδους. Δεν ξέρω αν χρειάζεται πραγματικά καινούργια νομοθεσία, καινούργιες πρωτοβουλίες. Απλά νομίζω ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι ήδη υφιστάμενες ρυθμίσεις, οι ήδη υφιστάμενες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για την παρουσίαση, για την εργασία σας, για την απάντηση των ερωτήσεων, αλλά ξέχασα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε να λάβετε το λόγο. Μάσιμο Σαπιέρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Εξ όνομα τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα μάλιστα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο ειλικρινά για την πρωτοβουλία του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει την έκθεση και τα βασικά ευρήματα και συμπεράσματά της. Επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ σε τρία θέματα. Υπάρχει ισχυρή σύγκληση μεταξύ της σημενής δραστηριότητας και πρωτοβουλειών ε, σε κοινοτικό επίπεδο ε, και σε επίπεδο κρατομελών και τις ε, απόψεις οποίες καταλήγει η έκθεση. Πέρυσι είχαμε αυτή την εταιρική σχέση για τη συνεργασία μεταξύ ερευνητών και πραγματικά τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν αυτά τα προγράμματα μέσω εθνικών προγραμμάτων και ελπίζουμε τις ερχόμενες εβδομάδες τα περισσότερα κράτη να έχουν εγκρίνει τα σχετικά προγράμματα. Το δεύτερο αφορά την κοινωνική ασφάλιση και ε, δικαιώματα για συμπληρωματική σύνταξη. Συνεργαζόμαστε πάλι με τα κράτη-μέλη και θα ήθελα να σας θυμίσω, μου επιτρέπετε, ότι το Μάιο του 2009 το Συμβούλιο, αν θυμάμαι καλά, Ο Ισπανός ε, Υπουργός ε, Έρευνας ε, έκανε μία πρόταση να γίνει ένα κοινό συμβούλιο με την ανταγωνιστικότητα και την ΕΠΣΚΟ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για τη θετική αξιολόγηση της πρωτοβουλίας ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφέρω μόνο τον Ευρωπαϊκό Χάρτη που είναι ορόσημο και ακρογωνίως λίθος και ε, ξεκίνησαμε και ένα μηχανισμό πριν από λίγους μήνες για τη στρατηγική ε, ανθρωπίνων πόρων για τους ερευνητές. Μπορεί να το βρείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα για να μεταφραστεί στην πράξη ο χάρτης αυτός στη ζωή των θεσμικών οργάνων. Και τέλος, Βεβαίω, θέλουμε να έχουμε συλλογή στατιστικών στοιχείων. Πολλές δραστηριότητες και δράσεις ε, αναλαμβάνουμε και τελειώνω λέγοντας ότι προσβλέπουμε να έχουμε και άλλε ευκαιρίες να συναντηθούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις ε, και σκέψεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται και αυτό το θέμα στη Μέση Διάταξη, λέει ο Για σήμερα βέβαια. Αλλά παρακαλώ και τη Γραμματεία να έχει υπόψη της ότι αυτά τα θέματα ερευνητικά θα πρέπει να τα συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος όπως είπαν και κάποιοι συνάδελφοι. Κοινή συζήτηση τώρα στο θέμα 5 και 6 είναι η φαρμακοεπαγρύπνηση. Περίπλοκη λέξη. Έχουμε κοινή συζήτηση λοιπόν και η συγγήτρια είναι η κυρία Μισελ Ριβαζή. Σωστά σας λέω, ελπίζω και σας δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήρθε στη σωστή στιγμή αυτή η έκθεση για την οδηγία, διότι αν δούμε τι συμβαίνει με τα φάρμακα και ιδιαίτερα με τις παρενέργειες, πρέπει να ενισχυθεί η επαγρύπνηση για προστασία του πολίτη. Έχουμε πολλά επίκαιρα πράγματα σχετικά με την νέα γρήπη. Γιατί πετράπει ένα φάρμακο με έγκριση δύο μηνών. Πήγει δηλαδή το θέμα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα εποπτείας υπεραποτελεσματικό. Έπειτα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολλά φάρμακα, το Vioxx που δημιούργησε επέφερε και θανάτους καρδιοκυκλοφορικά, η παροξετίνα, αντικαταθλιπτικά, το Προζάκ, αύξησαν τις αυτοκτονίες, το Ziprexac, αύξησε το διαβήτη και τα προβλήματα του μεταβολισμού. Έπειτα ε, έχουμε όλο και περισσότερες παρενέργειες που τελικά τα πληρώνει το κοινωνικό σύνολο. 5% ε, αύξηση των ημερών στα νοσοκομεία, 5% αύξηση των θανάτων μέσα στα νοσοκομεία λόγω ακριβώς αυτών των παρενεργειών. Οι νέες προτάσεις της Κομισιόν είναι πρόοδος και σημαντική μάλιστα σε σχέση με τις 10 Δεκεμβρίου του 2008 αλλά παραμένουν επαρκείς για να ενισχυθεί η φαρμακοεπαγρύπνηση στην Ευρώπη. μια ε, έγκριση στο να μπει σε εμπορία ένα φάρμακο θα πρέπει να στηρίζει σε πολλές κλινικές μελέτες, έρευνες με πολλά δείγματα και να υπάρχει και εποπτεία και πληροφόρηση. Είναι σημαντικό να πάρουμε τμήματα της οδηγίας και να τα βελτιώσουμε. Πρόβλημα υπάρχει εκεί που έχουμε τη διαχείριση του κινδύνου. Διότι αν πετύχουμε καλύτερη διαχείριση, αν αυξηθεί μάλλον ο κίνδυνος, τότε θα υπάρχει κίνδυνος αν μπει πρόωρα στην εμπορία ένα φάρμακο. Τι εννοώ. Ένα φάρμακο πριν μπει στο εμπόριο πρέπει να ε, αποτελέσει αντικείμενο έρευνα με συγκεκριμένα δείγματα και η φαρμακοεπαγρύπνηση σημαίνει να έχουμε λιγότερε παρενέργειες, να έχουμε λιγότερη ζημιά στον πληθυσμό γενικότερα. Η πρόταση τη Κομισιόν προβλέπει γενίκευση της δυνατότητας ε, προγραμμάτων διαχείριση του κινδύνου, πιο συγκεκριμένα όταν υπάρχουν ανησυχίε σχετικά με αρνητικέ εξελίξεις, σχέση ωφέλου κινδύνου του συγκεκριμένου φαρμάκου που να είναι αναλογικό, ανάλογο μάλλον με τον κίνδυνο. Η εμπειρία μας δείχνει ότι τα προγράμματα διαχείρισης του κινδύνου συχνά χρησιμοποιούνται για να καθησυχαστεί το κοινό όταν πρόκειται πρόωρα να μπει στην αγορά ένα προϊόν το οποίο η αξιολόγηση είναι ανεπαρκής. Να σας δώσω και παραδείγματα. Ρίμονταμπο ή το Σαμπίξ ή και άλλα που δόθηκαν πολύ γρήγορα οι εγκρίσεις λέγοντας θα γίνουν, ε, ε, υπάρχουν, μάλλον θα γίνουν έρευνες αργότερα. Δεύτερο πρόβλημα προς βελτίωση είναι το πέρας της χρηματοδότησης της, εκ μέρους του δημοσίου δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης. Έτσι μειώνεται η φαρμακοεπαγρύπνηση σε παρόχους ε, φαρμακευτικών υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή αν υπάρχει η υποχρέωση το δημόσιο να παρεμβαίνει δημιουργείται και αυτό το πρόβλημα. Τρίτο στοιχείο είναι η ενίσχυση του ελέγχου εκ μέρους των ιδιωτικών επιχειρήσεων ε, στην συλλογή και ερμηνεία των δεδομένων. Αυτό είναι ένα μείζον πρόβλημα, διότι θεωρούμε ότι το να δοθεί ευθύνη στις φαρμακευτικές βιομηχανίες δίνοντάς στην αρμοδιότητα να συλλέγουν και να ερμηνεύουν τα στοιχεία, νομίζουμε ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα. Ακριβώ το αντίθετο. Εδώ έχουμε σύγκρουση συμφερόντων, διότι αν ζητήσετε από ένα εργαστήριο να συλλέξει πληροφορίε, να ερμηνεύσει πληροφορίε για ένα φάρμακο που το ίδιο το εργαστήριο παρασκεύασε, Φυσικά θα προτιμήσει το οικονομικό του συμφέρον και όχι το συμφέρον της υγείας του κοινού. Τέταρτο, η Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείριση των Κινδύνων. Χωρίς έγκριση, χωρίς αυτονομία η Επιτροπή αυτή. Γιατί να συσταθεί ένα νέο όργανο αν δεν είναι αυτόνομο και αν είναι απλώς συμβουλευτικό. Καλύτερα θα ήταν ε, να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης που θα συνεργάζεται με τα εθνικά συστήματα και που ιεραρχικά και διανοητικά, ας το πούμε, θα ήταν ανεξάρτητο από την, από την Επιτροπή. Διότι κάποιος που έδωσε την έγκριση να μπει στην αγορά ένα φάρμακο και είναι και στην Επιτροπή, τι θα πει, θα πει μετά ότι κακός έγινε αφού ο ίδιος έδωσε την έγκριση. Πέμπτο, η διάχυση των πληροφοριών σε μια μέγα βάση, έδρα βιζιλάνς όπως το λέμε, αυτό δημιουργεί το εξή πρόβλημα. Αυτή η βάση στοιχείων θα είναι προσβάσιμη, όπως είπε η Κομισιόν, μόνο για τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Από αυτούς μόνο θα είναι προσπελάσιμη. Ποιες είναι αυτές οι αρχές όμως. Και γιατί αυτή η τεράστια βάση δεδομένων να μην είναι προσπελάσιμη και από ανεξάρτητους δεν μπορώ να κάνω μια αξιολόγηση των παρενεργειών φαρμάκων. Ξέρω ότι στην Ευρώπη είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι σε θέματα διαφάνεια. Εδώ δεν έχουμε διαφάνεια. Αν κάποιο έχει λόγους να, να ψάξει αυτέ τι πληροφορίες, γιατί να μην μπορεί. Έκτο, πρέπει να έχουμε ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Υπάρχει σε ορισμένε χώρες Υπάρχουν συστήματα, δημόσια συστήματα φαρμακοπαγρύπνησης. Η Κομισιόν δεν επιμένει ε, αρκετά στο να τα ενθαρρύνει. Και τέλος, αδιαφάνεια στα δεδομένα αν δεν υπάρχει πρόσβαση περιοδική ασφάλειας. Με το πρόσχημα ε, της, ε, του εμπορικού εμπιστευτικού χαρακτήρα των στοιχείων αυτών στη φαρμακοεπαγρύπνηση, επιβάλλεται να υπάρχει πρόσβαση στις εκθέσεις αυτές και στις εκθέσεις αξιολόγησης. Πρέπει όλα αυτά να δημοσιεύονται. Και τελειώνω με το εξή. Η ομάδα μας θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθούν τα κριτήρια εκχώρησης ενός πιο ασφαλούς φαρμάκου και άδεια. Πρέπει να υπάρχει ένα κριτήριο για να μπει το φάρμακο στην αγορά. Τα νέα φάρμακα να αποτελούν πρόοδο στη θεραπεία και να μην υπάρχουν παρενέργειες για το κοινό. Διότι αν δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία για το νέο φάρμακο, γιατί να δοθεί έγκριση. Αν πρόκειται να δημιουργήσει παρενέργειες. Οι αρχές πρέπει να μπορούν να είναι ανεξάρτητες ως προς τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητες και οικονομικά και στο ερευνητικό σκέλος και να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ανάφερα σε αυτό πριν και για του εμπεριογνώμονες και για αυτού οι οποίοι θα αποτελούν μέλη αυτή τη Ευρωπαϊκό, αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μάλλον. Τέλος ενίσχυση της διαφάνειας ω προ τον ασθενή να μπορεί να ξέρει το προφίλ των παρενεργειών, να είναι γραμμένο αυτό μέσα στο κουτί και με μεγάλα γράμματα να προσοχή, το φάρμακο αυτό δεν είχε τα, πρωτόκολλα, το, τα κριτήρια πρωτοκόλλου ανάπτυξης για τόσα χρόνια όπως απαιτείται, να ειδοποιείται δηλαδή ο ασθενής να ξέρει. Πρέπει να κάνουμε πολλέ τροπολογίε. Αλλά είναι μεγάλη ευκαιρία. Πρέπει να βελτιωθεί αυτή η οδηγία, διότι αν την αφήσουμε έτσι όπως είναι, δεν απαντάει στα κοινωνικά αιτήματα. Ευχαριστώ. Α, δεν είχα ανοίξει μικρόφωνο. Λοιπόν, σκιώδης ηγητής, κύριος Κορέρα Τεκάμπος πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ε, ευχαριστώ και πρέπει να σας πω ότι η ομάδα μας συμφωνεί με πολλά από τα συμπεράσματα της εισηγητρίας διότι κατανοούμε ότι τα προ... Ε, γράμματα, μάλλον οι πρόοδοι που έχουν γίνει στη θητεία αυτή είναι καλές αλλά ανεπαρκείς. Θα πρέπει να κοιτάξουμε αυτή τη σχέση κόστους-οφέλειας αλλά και ποιος πληρώνει το κόστος. Τρεις είναι οι εναλλακτικέ λύσεις. Ο καταναλωτής, τα κράτη-μέλη ή επιχειρήσεις. Μέχρι τώρα το κόστος επιβαρύνει κυρίως τον καταναλωτή, τον άρρωστο, ούτε τα κράτη-μέλη, ούτε τους φαρμακοβιομηχάνους. Αυτή το πολύ πολύ να υφίσταται τις συνέπειες των ε, διενέξεων των νομικών που πάντα έχουν αβέβαιο αποτέλεσμα. Για να έχουμε λοιπόν καλύτερη πρόληψη εδώ θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Το σύστημα διαχείρισης κινδύνου που προτείνεται με ΑΙ είναι ε, ε, χρήσιμο για την ενημέρωση ως προς τον κίνδυνο και για την αποτροπή αλλά δεν έρχεται να καταργήσει τον κίνδυνο. Και είναι γεγονός επίσης ότι το σύστημα αυτό που προτείνεται ε, απλουστεύει τα σημειώματα για τις αντενδείξεις και τις παρενέργειες και αυτό είναι θετικό. Επίσης, οι ρυθμιστικοί οργανισμοί τύπου ΕΟΦ ε, που θα πρέπει να ενημερώνουν ε, την ε, πληροφόρηση και την τεκμηρίωση για τους ιατρικούς κινδύνους. Όλα αυτά είναι ωραία και καλά. Αλλά δεν αρκεί η παρακολούθηση, η επαγρύπνηση. Θα πρέπει να βγάζουμε και συμπεράσματα ή να απαιτούμε απάντηση από κάποιον που έχει πάρει άδεια κυκλοφορίας ε, του φαρμάκου στην αγορά. Οι εκθέσει ασφαλείας κάνουν μια διάκριση ανάμεσα σε φάρμακα χαμηλού κινδύνου και συμφωνώ ότι το φάρμακο χαμηλού κινδύνου δεν θα πρέπει να έχει τις ίδιες απαιτήσει με εκείνο το υψηλού κινδύνου. Αλλά στην πράξη νομίζω είναι πολύ δύσκολο να ε, κάνει κανείς τη διάκριση αυτή. Η συγκήτρια ανέφερε δύο φάρμακα, Βίοξ ε, και Προζάκ. Αυτό τι είναι, χαμηλού κινδύνου ή υψηλού. τουλάχιστον ένα από τα δύο από χέρι δεν θεωρείται υψηλού κινδύνου. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αμφισημία και θα πρέπει να ξεκαθαριστεί οπωσδήποτε. Καλή απλούστευση του συστήματος και η επικέντρωσή του. Η συγκέντρωση μάλλον. Για την δραστική ουσία. Είναι θετικό, λέει αυτό, για να αποφεύγονται, πώς να το πω, τα προβλήματα. Ε, εάν δεν αντιμετωπίζουμε τη δραστική ουσία γενικά με τον ίδιο τρόπο, μπορεί κάποιος παρασκευαστής να αδιαφορεί, να αγνοεί ε, τις συνέπειες χωρίς να υφίσταται κανένα ανέλεγχο και καμία επαλήθευση. Να υπάρχουν συνθήκες ε, για κάθε ενεργή δραστική ε, ουσία και αυτό να ελέγχεται από εκεί και πέρα. Τέλος, το σύστημα επαγρύπνησης έχει λειτουργήσει παρόλα αυτά για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Αλλά δεν ήταν αρκετά ισχυρό για να μπορέσει να επεκταθεί και στις περιπτώσεις που αναφέραμε. Τι λέμε λοιπόν τώρα. Θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για τον κίνδυνο και να ξέρουμε ποιες είναι οι πηγές που ενημερώνουν. Η πρόταση λοιπόν της Ήτρας λέγει ότι θα πρέπει να αναγράφεται στο συνοδευτικό σημείωμα μέσα στο φάρμακο ε, ε, η ύπαρξη παρενεργειών και ε, ανεπιθυμήτων ε, ενεργειών. Αυτό μας καλύπτει, μας στάνει ή θέλουμε να υπάρχει όσο γίνεται μεγαλύτερη δυνατή πληροφόρηση και από άλλες πηγές. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σπάλτσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς πρέπει να πω ότι η φαρμακοεπαγρύπνηση είναι για μένα μια έννοια που άκουσα σήμερα για πρώτη φορά στη ζωή μου, διαβάζοντας την έκθεση. Εγώ ήξερα για παρενέργειες, για ανεπιθύμητες ενέργειες, πρώτη φορά βλέπω φαρμακοεπαγρύπνηση. Εν ε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Η κυρία Ριβασί αναρωτήθηκε και η ίδια ε, για κάτι που με προβληματίζει και εμένα. Μίλησε για τους κινδύνους. Και αναφέρθηκε σε μια νέα επιστημονική επιτροπή ή επιστημονικό συμβούλιο για τη φαρμακοεπαγρύπνηση και ότι θα παίξει σημαντικότατο ρόλο. Εμείς τώρα γιατί είμαστε αρμόδιοι για αυτή την έκθεση και γιατί όχι Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού πρόκειται για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Από πού και ως πού είμαστε εμείς αρμόδιοι, γιατί είναι και φάρμακα. Η βιομηχανία φαρμάκων είναι η δεύτερη σημαντικότερη βιομηχανία, σύμφωνα με τη γνώμη ορισμένων, μετά τη βιομηχανία ε, οπλικών συστημάτων και οι άρρωστοι είναι άνθρωποι ακριβώς ασθενείς και εξασθενημένοι που είναι εκτεθειμένοι στα νύχια αυτών των φαρμακευτικών εταιριών που έχουν και πάρα πολύ ισχυρό λόμπι. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Οι φαρμακευτικές εταιρείε έχουν πάρα πολύ ισχυρά λόμπι. Εμείς πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι ένα τέτοιο συμβούλιο ή μια τέτοια επιτροπή θα είναι ανεξάρτητη. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι πολύ κρίσιμο αυτό. Και μετά, βάση δεδομένων. Γιατί να είναι περιορισμένη η πρόσβαση, για να μην, να μην είναι προσπελάσιμη αυτή η βάση δεδομένων σε ανεξάρτητους ερευνητές και επιστήμονες. Ευχαριστώ. Προσπαθώ να σας απαντήσω για το ποιος είναι αρμόδιος. Εμείς γνωμοδοτούμε. Opinion λέει εδώ. Καθήλυνα αρμόδια είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος, όπως είπατε κι εσείς. Εμείς λέμε τη γνώμη μας. Γνωμοδότηση λέγεται αυτό. Γι' αυτό πρέπει και να το συζητάμε. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιο είναι η κυρία Σάντσες. Έχετε το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ και καλησπέρα σας. Όντω, με δυναμική αυτή πρόταση, αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι το εξή, να βελτιώσουμε το σύστημα φαρμακοϊπαγρύπνηση. Αυτό έχει λειτουργήσει, δεν θα πρέπει να πανικοβαλόμαστε για το παρελθόν. Επειδή υποβλήθηκε μια πρόταση βελτίωσης του συστήματος, έχουμε περιθώριο βελτίωση και μάλιστα μεγάλο ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την καλύτερη χρήση των πόρων, σε ό,τι αφορά το δίκτυο των αρχών, για να επικεντρωθούμε δηλαδή σε σημαντικά θέματα ασφάλειας μετά από την έγκριση των φαρμάκων. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Να απαντήσω σε κάποια από τα ερωτήματα και στα σχόλια που έγιναν, για να εξηγήσω ποια ήταν η πρόθεσή μας με την πρόταση αυτή. Ήταν η πρόθεσή μας να βελτιώσουμε την ε, εποπτεία μετά τη θέση στην εμπορία των φαρμάκων. Όχι όμως σε καμία περίπτωση εις βάρος. Όχι ότι θα ε, χαλαρώσουμε τους κανόνες για την έγκριση για θέση στην αγορά. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει. Και δεν θα διαβρύνουμε τις εξαιρέσεις όπου δίδεται έγκριση προτού έχουν γίνει προκλινικές και κλινικές ε, δοκιμές. Όπως για παράδειγμα, σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την κατηγορία υπάρχει και το παράδειγμα της, ε, του εμβολίου κατά της γρήπης, της πανδημικής γρήπης. Χρειάζεται λοιπόν ε, μια πλήρης αξιολόγηση των κινδύνων. Αυτό δυστυχώς δεν σημαίνει ότι τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά δεν έχουν κανένα απόλυτος κίνδυνο, δυστυχώς. Και δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να δοκιμαστεί το φάρμακο σε μεγάλο ε, δείγμα πληθυσμού. Πολύ μεγαλύτερο από, το, από την κλινική δοκιμή. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τα φάρμακα και πώς αντιδρούν στην πραγματική ζωή και να συνεχίσει η αξιολόγησή τους. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να διευκρινιστεί στο κείμενο περί έγκρισης ε, για κυκλοφορία στην αγορά. Ευχαρίστως να συνεχίσουμε τη συζήτηση, ε, για το θέμα αυτό. Το θέμα της ανεξαρτησίας ε, το έθεσαν πολλοί ομιλητές. Πώς εγγυόμαστε την ανεξαρτησία όταν επιβάλλουμε έξοδα η κατάσταση πώς έχει. Οι πιο πολλές αρμόδιες αρχές έχουν την δυνατότητα να επενδύσουν στη φάση πριν τεθεί στην αγορά και μετά αφού έχει τεθεί στην αγορά το φάρμακο. Όταν η ε, πόροι αυτή βρίσκονται υπό τον έλεγχο των δημόσιων αρχών. Υπάρχει ανεξαρτησία φυσικά. Επίσης ε, τέθηκε το θέμα της ανεξαρτησίας της ε, Επιτροπής από την βιομηχανία και από τις δημόσιες ε, αρχές. Ήδη έχουμε πολλές επιτροπές που λειτουργούν σε ό,τι αφορά το κοινωτικό πλαίσιο για τα φάρμακα και παραδοσιακά απαρτίζονται από εμπειρογνώμονες από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Νομίζω ότι έχουμε ένα αρκετά αξιόπιστο σύστημα σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία από τη βιομηχανία. Είναι δυνατό αυτό, παρά το προφανές ε, γεγονός ότι πρόκειται για ένα σημαντικό τμήμα της βιομηχανίας. Ωστόσο, στην παρούσα πρόταση προτείνουμε το εξή. Προτείνουμε μια ελαφρώς τροποποιημένη σύνθεση για την ε, Επιτροπή αυτό που με οδηγεί στα σχόλια της κυρίας Ριβάση. Δεν προτείνουμε η Επιτροπή αυτή να έχει εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, όπως οι προηγούμενες επιτροπές στο Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τα Φάρμακα, αλλά προτείνουμε μια πραγματική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, όπου θα χρησιμοποιούμε και τους πόρους από τις εθνικές αρχές και από τις εθνικές αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και από τις ε, οργανώσεις εμπειρογνωμόνων. Γι' αυτό λοιπόν ε, διοργανώσαμε ένα δημόσιο διαγωνισμό εκδήλωση ενδιαφέροντος. Τέλος, να σημειώσω κάτι σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια. Προσπαθήσαμε ιδιαίτερα να προωθήσουμε τα θέματα διαφάνειας σε αυτή την πρόταση με διάφορα μέτρα. Ε, στο σελίδες, ε, κόμβι στο ίντερνετ κτλ. Και η διαφάνεια αποτελεί ε, μία, έναν από τους στόχους της πρότασης αυτής. Σε ό,τι αφορά την βάση δεδομένων, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι τα στοιχεία της φαρμακοεπαγρύπνησης αποτελούν όλες, αποτελούνται από όλες τις ε, παρενέργειες των φαρμάκων σε όλη την αγορά. Το θέμα δεν είναι να προστατεύσουμε το εμπορικό απόρριτο. Το θέμα είναι να προστατεύσουμε προσωπικά δεδομένα. Γι' αυτό αυτό που λέμε στην πρόταση είναι το εξή. Να υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση για το κοινό για να προστατευτεί η ανωνυμία των ατόμων στα οποία έχουν σημειωθεί ανταντήξεις παρενέργειες. Αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά την πτυχή της διαφάνειας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Σαφέστατη η απάντηση. Νομίζω ότι μπορούμε έτσι να κλείσουμε το 5 και το 6, να περάσουμε στο 6 και 7 λέει ο πρόεδρο, μάλιστα 7 και στο 8. Ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Και εδώ κοινή συζήτηση. Και να δώσω το λόγο στον κύριο Χατζημαρκάκη, που είναι ο εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που είστε ακόμα εδώ 5,5 ε, ώρα, πέμπτη απόγευμα. Και εγώ χαίρομαι που σα βλέπω. Και αν τα πείτε γρήγορα θα φύγουμε και γρήγορα. Ωραία, γρήγορα θα τα πω. Αυτά τα δύο θέματα είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ του Στο σημείο 7 είναι η πανευρωπαϊκή Ένα κώδικα για την ενημέρωση των ασθενών και ε, πρόκειται για φάρμακα αποκλειστικά ε, υποχρεωτική συνταγογράφηση. Το σημείο 8 είναι κανονισμός που αφορά περισσότερο ε, θέματα ενημέρωσης του κοινού πάλι για, για φάρμακα υποχρεωτικής συνταγογράφησης. Το θέμα είναι εκρηκτικό πολιτικά και πολύ καυτό γενικότερα και δυστυχώς το πρίσμα στη συζήτηση μέχρι τώρα ήταν ως εξής και το λέω ευθύ εξ αρχή, ότι πρόκειται κυρίως, λέει, για διαφήμιση. Αυτό είναι εσφαλμένο και ψευδές. Πρόκειται για ενημέρωση. Οι πολίτε οι ασθενεί έχουν δικαίωμα να είναι επαρκώς ενημερωμένοι και για τις ασθένειες και για τα φάρμακα. Σε τελική ανάλυση πρόκειται για δικαιώματα των ασθενών. Ε, Επισημένω στους συναδέλφους ότι το θέμα αυτό το έχουμε ήδη συζητήσει και να βάγισε το 2003 στο Κοινοβούλιο και παρακαλώ να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά σας παραπέμπω και στο εξή. Η Σουηδική Προεδρία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος είπε ήδη ότι παρόλο που ως παράδειγμα έχει το σουηδικό μοντέλο δεν θέλει να το φέρει πολύ στο σκήνιο κατά τη διάρκεια της δική της ε, προεδρίας γιατί δεν έχει τις απαραίτητες πλειοψηφίες προφανώς. Περί τίνος πρόκειται. Οι ασθενείς, οι καταναλωτές ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για την ίδια τους την υγεία και ακόμα ε, περισσότερο για τη θεραπεία και την πρόληψη ε, των ασθενειών τους και θέλουν να έχουν και γνώμη. Η βέλτιστη όμως αντιμετώπιση είναι δυνατή μόνο εφόσον γνωρίζουν πραγματικά οι ασθενείς τι φάρμακα παίρνουν και να μην επαφίενται μόνο στο γιατρό τους, να είναι υποχρεωμένοι κιόλα να το κάνουν. Θα πρέπει να λαμβάνουν μια ε, ενημερωμένη απόφαση και αυτό έχει και στοιχεία πρόληψης, διότι ε, ασθενείς που έχουν πιο μακροπρόθεσμη προοπτική μειώνουν το κόστος για την κοινωνική ασφάλιση, αρρωσταίνουν πιο σπάνια, αρρωσταίνουν λίγο και επειδή είναι ενημερωμένοι και ε, συνειδητοί και γνώση τους συμβαίνουν όλα αυτά, μειώνεται το κόστος για την υγεία. Αλλά θα πρέπει να είναι ε, τα στοιχεία κατανοητά, αντικειμενικά και χωρίς διαφήμιση. Και όχι μόνο μέσω των γιατρών, αλλά και με άμεση πληροφόρηση. Ερώτηση, πώς θα γίνουν όλα αυτά. Να περιμένουμε δηλαδή να αρρωστήσει κάποιος. Είναι ο μηχανισμός πους δηλαδή ε, ε, παίρνει τις πληροφορίες που συμβαίνει κατά κανόνα. Εμείς είμαστε πολύ προσεκτικοί Και προβλέπει και ο κανονισμός να υπάρχουν, ε, αυτό το προηγούμενο που σας είπα λέγεται ο μηχανισμός pull εκ των υστέρων. Τώρα υπάρχει ο μηχανισμός push, δηλαδή να οθούνται, να ενημερώνονται με ε, πληροφορίες ε, που φτάνουν σε αυτούς οι ασθενείς. Πώς φτάνουν οι πληροφορίες σε αυτούς. Μέχρι τώρα, ε, με το σημείωμα που υπάρχει μέσα στο φάρμακο, ο καθένας από εσά γνωρίζει ότι αν πάρετε ένα φάρμακο και διαβάσετε ε, το σημείωμα είναι κατανόητο. Τραπεζομάντιλα είναι, ε, να και αγχώνουν μάλιστα τους ασθενείς. Άμα κάτσω και διαβάσω τι γράφει αυτό το χαρτάκι, κάηκα. Δεν <laughs> θέλω μετά να πάρω και το φάρμακο. Ε, πρόκειται λοιπόν για πληροφόρηση που έχει ε, γραφτεί από νομικούς για νομικούς. Και η μαμά μας πούμε δεν το καταλαβαίνει αυτό το χαρτάκι. Επίσης, έτσι ναι, Εγώ καμιά φορά δεν τα διαβάζω και δεν είμαι και νομικό. Τι, να κάνει και η μάνα μου. Λοιπόν, η πληροφόρηση εξαρτάται Επίση, και κατά πόσο και πόσο καλά μπορεί ο καθένα να χειρίζεται το ίντερνετ. Γιατί πολλοί και περισσότεροι πολίτε πηγαίνουν στο διαδίκτυο και παίρνουν ενημέρωση. Αλλά εδώ έχουμε μία ανισότητα. Διότι τα περισσότερα στοιχεία που αφορούν φάρμακα είναι στα αγγλικά. Και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Πρώτον, Δηλαδή κάποιο Λετωνός που δεν ξέρει αγγλικά τι θα κάνει ο άνθρωπος. Δεν έχει την ίδια πρόσβαση. Επιπλέον, έχουμε και ψευδή στοιχεία. Ε, μη αξιόπιστα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχουμε ανταγωνιστές που διαδίδουν ψευδή στοιχεία και πληροφορίε για άλλα φάρμακα. Είναι κακό πράγμα αυτό. Άρα χρειάζεται πιστοποιημένη, αξιόπιστη ενημέρωση και σελίδες, στο διαδίκτυο. Και γι' αυτό λέει κάποια πράγματα η πρόταση. Επιπλέον θα πρέπει να σκεφτούμε ότι βέβαια εκτό από το χαρτάκι μέσα στο φάρμακο παίζει ρόλο και ο γιατρός που το συνταγογραφεί βεβαίω, αλλά κατά μέσο όρο η διάρκεια μιας επίσκεψης στο γιατρό είναι ένα τέταρτο το τρίμηνο σε όλη την Ευρώπη. Ένα τέταρτο διαθέτει ο κάθε γιατρός στον ασθενή του το τρίμηνο. Φανταστείτε τώρα τι χρονικό διάστημα είναι αυτό. Άρα θα πρέπει ο ίδιος ο ασθενής να πάει να το ψάξει. Και Τελικά θα πρέπει να παίρνει την απόφαση ο γιατρός. Προφανώς παίζει εκείνο τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά σιγά σιγά να συμμετέχει όλο και περισσότερο ασθενής. Τώρα, τι καλωσορίζουμε σε αυτή την πρόταση. είναι γνωμοδότηση για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, είναι ένα ενισχυμένο σημείωμα μέσα στο φάρμακο, που είναι το α και το ω ε, της πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει επιτέλους να γίνει εύληπτο αυτό το χαρτάκι, κατανοητό για τον ασθενή. Στη Γερμανία, που είναι η πατρίδα μου και δεν ξέρω καλύτερα από τις άλλες χώρες, αυτό είναι ε, ε, υποχρεωτικό διανόμου. Αλλά διανόμου υποχρεωτικό δεν σημαίνει ότι το καταλαβαίνει και ο ασθενή τελικά όταν το διαβάζει. Λοιπόν, καλύτερη ενημέρωση, εκτενέστερη, ε, ειδικότερη για την ασθένεια του καθενό και όλα αυτά να γίνουν με τρόπο ελκυστικό για τον ασθενή. Ε, δεν είναι και υπερβολικά αυτά που ζητάμε. Διότι τελικά στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί αυτών πρόκειται. Και επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται για διαφήμιση, η οποία ρητός αποκλείεται. Άκουσα αυτή τη βδομάδα ότι συνεδριάζει το φόρουμ το φαρμακευτικό υψηλού επίπεδου. 12 κριτήρια έχουμε βάλει ποιοτικά, ε, χρόνια ολόκληρα που συνεδριάζουμε, για να διαχωριστεί η διαφήμιση από την ενημέρωση. Και παρακαλώ να μην ε, πέσουν οι συνάδελφοι στην παγίδα ορισμένων ε, ομάδων που ασκούν πίεση. Δεν θέλει η βιομηχανία να κάνει διαφήμιση. δεν θέλουν ούτε καν οι φαρμακευτικές εταιρείες να κάνουν διαφήμιση. Και σας λέω κάτι που λένε και οι ορισμένοι φορείς κοινωνικής ε, ασφάλισης. Και αυτό είναι παραπλανητικό, διότι λέει ότι θα πρέπει αυτή η πρόταση να απορριφθεί για το καλό ε, του ασθενούς. Γιατί αυτοί φοβούνται το υψηλότερο κόστος. Μα δεν έχουμε υψηλότερο κόστο. Όταν ο πολίτη γνωρίζει περισσότερα, δρά προληπτικά, αρρωσταίνει λιγότερο και μειώνεται το κόστο για τι ε, ασφαλιστικές εταιρείες και τα ταμεία. Τελικά, λοιπόν, ενημέρωση είναι ένα πρώτο βήμα. Στην ΕΜΕΑ, στο φορέα στο Λονδίνο, έχουμε έγκριση για 400 φάρμακα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτή η agency υπηρεσία για τα φάρμακα ε, έχει εγκρίνει 400 έχουν κάποια κονδύλια που δεν τους φτάνουν και θα πρέπει να αυξηθούν γιατί δεν θα μπορέσουν να το κάνουν χρειάζεται και κάποια ταχύτητα αυτό. Τώρα, τα υπόλοιπα φάρμακα που θα πρέπει να εγκριθούν από τις εθνικές ε, υπηρεσίες, το ΝΕΟΦ, ε, επίσης θα έχουν τέτοια ενημερωτικά σημεία. Σε όλα τα κράτη δεν είναι εύκολο να υπάρχει έλεγχος εκ των προτέρων, εξάντε, για τη Σουηδία για παράδειγμα, ισχύει αυτό ε, και για τις χώρες αυτές επιτρέπονται εξαιρέσεις. Να μην έχουμε εκ των προτέρων έλεγχο. Ο εκ των υστέρων έλεγχος της πληροφόρηση είναι έτσι και ω καλύτερο γιατί είναι λιγότερο γραφειοκρατικό και αποτελεσματικός, αλλά θα πρέπει να είναι υψηλό το πρόστιμο σε περίπτωση παράβασης. Στη Σουηδία είναι χαμηλό και η εμπειρία λέει ότι θα πρέπει να αυξηθεί το πρόστιμο και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εκεί χρειάζεται βελτίωση, πρόταση να έχουμε ενιαίες κυρώσεις για να έχουν και αποτρεπτικό χαρακτήρα, αλλιώς δεν βοηθάει τίποτα. Και χρειάζεται επίση αναρμόνιση του ορισμού των δημοσιεύσεων που σχετίζονται με την υγεία. Παράδειγμα, ανοίξει ένα περιοδικό και αν υπάρχει τέτοια ενημέρωση, να υπάρχει ενιαία σχήμα, ενιαία μορφή για να καταλαβαίνει ο ασθενή, αλλιώ θα νομίζει ότι είναι διαφήμιση. Αυτό να ε, οριστεί σαφώς και ενιαία. Τώρα, οι πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου συζήτησαν αυτό το θέμα γιατί συναντήθηκα με τους σκιώδης και θέλουμε να γίνει ακρόαση, hearing, όχι από την Επιτροπή μας αλλά από τις πολιτικές ομάδες για να μην σας επιβαρύνουμε κύριε Πρόεδρε. Ωστόσο, Χρειάζεται να γίνει τέτοια κρόαση, υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα. Να σας ενημερώσω για το χρονοδιάγραμμα, διότι αναβλήθηκε η αρχική ημερομηνία ε, στην καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος θα γίνει ψηφοφορία μόλις τον Απρίλιο και μετά το Μάιο στην Ολομέλεια. Γι' αυτό στο Δεκέμβριο, οπότε να το βρω. Στις 12 Νοεμβρίου, συγγνώμη, θα πάρετε την πρόταση για την έκθεση μέσω του εισηγητού. Στις 3 Δεκεμβρίου θα ε, ξανασυζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή μας και στις 9 Δεκεμβρίου λίγη η προθεσμία ε, για την κατάθεση των τροπολογιών σας, αλλά καλά, μην μας κατακλείσετε και με τροπολογίες για να ε, στείλουμε γρήγορα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος τη νομοδότησή μας. Είναι πάρα πολύ συνεργάσιμοι οι συνάδελφοι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, οι περισσότεροι τουλάχιστον και θα μας ακολουθήσουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Έμαθα πολλά από αυτά που μας είπατε σε τέτοιες λεπτομέρειε και επιτρέψτε μου αυτό το αστείακι τέτοιες ώρες ότι το σημαντικότερο είναι ότι η μαμά σα θα μπορεί να διαβάζει και τα χαρτάκια στα φάρμακα στο μέλλον και είναι πάρα πολύ σημαντικό επιχείρημα και να το χωνέψουμε όλοι και να βάλουμε τα δυνατά μα για να πετύχει. Ο Σκιώδη, συζητητής των σοσιαλιστών έχει το λόγο τώρα και ο Σκορέρα Ντεκάμπος. Eh, e και εγώ έμαθα πολλά. Πολύ ενδιαφέρουσα η εισαγωγή αυτή. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και θα περάσω κατευθείαν στις ερωτήσεις μου. Έχω κάποιες αντιφατικές πληροφορίες. Θα φαίνεται ότι η Σουηδική Προεδρία σκοπεύει να κινήσει μια νέα θέση για το πακέτο αυτό πριν το τέλος του εξαμήνου της. Η Σουηδική Προεδρία δεν φαίνεται να θέλει να συζητηθεί το πακέτο αυτό ή τουλάχιστον αυτά τα δύο κείμενα. Θα μπορούσε κάποιος να μου ξεκαθαρίσει τι ακριβώς σημαίνει. Τι ακριβώς σημαίνει. Το θέμα κλειδί εδώ είναι πληροφόρηση. Πληροφόρηση σε αντιδιαστολή με τη διαφήμιση. Μπορεί να παράξει κανείς, ε, να πολύ χρήσιμη πληροφορία, αλλά υπάρχει κίνδυνος αν παραέχουμε πολλές πληροφορίες. Και η πληροφορία αυτή σε μεγάλη ποσότητα πολλές φορές έρχεται μέσα στα σπίτια μας, μέσω των υπολογιστών και πολλές φορές είναι λάθος πληροφορία και επηρεαζόμαστε από αυτή την πληροφορία. Είναι πρόοδος αυτό στην κοινωνία. Πρέπει να γίνουν πολλές βελτιώσεις στο μέτωπο αυτό. Η βελτίωση της πληροφόρησης, η περίοδος των 60 ημερών πριν γίνει η σιωπηρή αποδοχή να δοθεί η πληροφορία και αν δεν υπάρξει αντίρρηση μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα τότε να θεωρείται εγκεκριμένη η πληροφορία έγκυρη. Αυτό πρέπει να βελτιωθεί το σύστημα. Όπως είπε ο εισηγητής, πρέπει να δούμε τι πήγε καλά, τι δουλεύει ως σύστημα. Έχει, ε, θα οργανωθεί μια ακρόαση. Καλώς. Θα μας βοηθήσει να δούμε τουλάχιστον σε δύο χώρες ποιες είναι οι βέλτιστες μέθοδοι. Πρέπει όμως κάπως να αλλάξουμε τις προθεσμίες για να το πετύχουμε αυτό. Να επεκτείνουμε τις προθεσμίες προς το μέλλον. Φυσικά συμφωνώ με αυτό το νομοθετικό κείμενο να ισχύει μόνο για φάρμακα που δίνονται με συνταγή. Άρα ο ρόλος του γιατρού, να δεν νομίζω ότι μόνο ο γιατρός θα πρέπει να έχει αυτή την πληροφορία, γιατί έχει και ασθενής. Και ασθενής θα πρέπει να πληροφορείται. Πρέπει να φροντίσουμε η πηγή της πληροφόρησης να είναι σωστή, η πληροφορία να είναι χρησιμοποιήσιμη. Υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν και να διορθωθούν. Δεν λέμε όχι. Δεν απορρίπτουμε αυτό το σχέδιο νομοθετήματος. Δεν θέλουμε να χαθεί η ευκαιρία να σημειωθεί η πρόοδος. Θέλουμε να ενισχυθούν και ρυθμιστικές εξουσίες όπου υπάρχουν. Ξέρουμε ότι υπάρχει δισταγμός εκ μέρους των ρυθμιστικών σωμάτων στα κράτη-μέλη στο να δεχτούν αυτές τις πληροφορίες. Τα επιχειρήματά τους δεν είναι πάντα αιτιολογημένα. Έλλειψη κονδυλίων λένε. Ή κατανάγκη θα υπάρξει ε, αύξηση του έργου και της γραφειοκρατίας Υπάρχουν επίσης και θέματα, υπάρχουν θέματα που θα μπορούσαν να ισχύσουν στην περίπτωση αυτή. Συμφωνώ με την εισηγητή ότι αν αλλάξουμε το χρονοδιάγραμμα πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να μα δοθεί χρόνο να αναλύσουμε το θέμα σε όλες τις λεπτομέρειε να δούμε τι διάφορε προοπτικέ που υπάρχουν. Ακόμα είμαστε στι πρώτε φάσει, στην επιφάνεια. Πρέπει να πάμε σε βάθο. αντικειμενικά όμω. και χωρί ε, να είμαστε προκατηλημένοι. Πρόεδρο. Κυρία Γκουτιέρης Κορτίνης, ε, καθυστέρησα, αλλά τα θέματα αυτά που μας τα βάζετε τελευταία μέρα, τελευταία ώρα, ε, να μην τα βάζει γραμματεία παρακαλώ τα σημαντικά θέματα τέτοιες ώρες. Συμφωνώ. Ε, γιατί συζήτησα με τον εισηγητή σχεδόν σε όλα. Θέλω να προσθέσω τα εξή. Πρώτον, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα δώσει καμία μελέτη και χαίρομαι πάρα πολύ που αναβάλλεται το χρονοδιάγραμμα έτσι και οι ημερομηνίε λίγο αλλάζουν. Γιατί έχουμε τόσους πολλούς στα επίγοντα αποδελτηριάσεις φαρμάκων στα νοσοκομεία. Το θέμα δεν είναι μόνο να έχει η βιομηχανία διαφάνεια, αλλά να αποφεύγουμε και τέτοια πράγματα. Ο κόσμος παίρνει λάθος φάρμακα και μετά τρέχει στα επίγοντα. Και ηλικιωμένοι που δεν θυμούνται τι έχουν πάρει κτλ., Θα μπορούσε ήδη ο φαρμακοποιός να μας δίνει τα φάρμακα μοιρασμένα σε κουτάκια, τι πρέπει να πάρουμε κάθε φορά λοιπά. Αυτό πολύ καλό θα ήταν. Λοιπόν, ο κόσμος παίρνει φάρμακα και πολλές φορές δεν τηρεάζεται για να μην σας πω ότι πάει και στον τάφο. Γιατί έχει αλλεργίες, έχει κάτι, να κατέβει τα φάρμακά του, δεν προσέχει. Είναι πολύ σημαντικό. Ε, συμφωνώ λοιπόν και για αυτά για τους γιατρούς και δεν είναι μόνο η μητέρα του φίλου Χατζημαρκάκη και εγώ θα μπορούσα να ήμουν η μητέρα του και δεν καταλαβαίνω αυτά που βλέπω όταν τα βλέπω και τα διαβάζω. Λοιπόν, στα προσπέκτους αυτά, στα φυλαδέκια θα πρέπει να είναι πολύ σύντομο ενημέρωση για αδαείς, όχι για τους ειδικού. Και να λέει μην ανακατεύετε το α φάρμακο με το β. Και αν έχετε αυτά τα συμπτώματα ή αν χάσετε βάρος, Δηλαδή όταν είσαι 40, ε, συγγνώμη, κιλά παραπάνω ή 40 λιγότερα δεν πρέπει να πάρεις την ίδια δόση. Με πολύ ε, χοντρά γράμματα και πολύ απλά πράγματα. Και κάτι ακόμα. Θα πρέπει να απαιτήσουμε στο διαδίκτυο να υπάρχει πιστοποίηση με σήμα, με ετικέτα ποιότητας. Και έτσι το ίδιο ε, ενημερωτικό υλικό που υπάρχει στο φυλάδιο να είναι και στο ίντερνετ, να μην έχουμε επιπλέον από το ίντερνετ και απ' έξω κάποιος να μπορεί να το ελέγχει. Και όχι μόνο αυτό, θα προτείνω και κάτι άλλο ακόμα παραπέρα. Προτείνω λοιπόν τα φάρμακα υψηλής κατανάλωσης να έχουν και προγράμματα τηλεφωνικά, να μας στέλνουμε SMS πώς να το πάρουμε το φάρμακό μας ένα ηλικιωμένο να μπορεί ας πούμε, με το τηλέφωνό του να βλέπει, να παίρνει ένα μήνυμα πώ θα πρέπει να, να παίρνει το κάθε φάρμακο. Να καταλάβει ο κόσμο, ακόμα και αν δεν θέλει, να μαθαίνει. Και αυτό είναι σημαντικό. Και αν η, ε, τα φαρμακεία τα δεχτούν όλα αυτά και μας βοηθούν, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Ε, έτσι και το κάνουν βέβαια τα φαρμακεία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια μικρή υπόδειξη. Καμιά φορά διερωτώμε Καμιά φορά διαρωτώμε ότι πολλά από αυτά που γράφουν τα σημειώματα αυτά και δεν τα καταλαβαίνουμε όλοι, αποφασίσαμε όλοι μαζί ότι πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι το λέω εμπαρόδο αυτό. Και καμιά φορά λέμε τι άλλο να μπει μετά στο σημείωμα και ερχόμαστε να απορούμε που δεν το καταλαβαίνει η ψυχή. Αυτά. Καλά που το αναφέραμε και αυτό. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Ερεν Σάντσες έχει το λόγο. Και μετά ο για να κλείσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ σύντομη. Γιατί ο κ. Κατζημαρκάκη εξήγησε τα προβλήματα και εξήγησε γιατί πρέπει να δράσουμε. Να σχολιάσω όμως κάποιες από τις παρατηρήσεις του. Καταρχάς, να πω ότι αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε με την πρόταση αυτή είναι να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο που θα μας επιτρέψει να παρέχουμε πληροφορίες οι οποίες γενικώ ζητούνται από την κοινωνία, από τους καταναλωτές, από τους ασθενείς. Ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσουμε την απαγόρευση της διαφήμισης. Άρα, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να θέσουμε σαφείς κανόνες για το ποιες πληροφορίες μπορούν να χορηγούνται και πώς μπορούν να χορηγούνται. Με όλες τις λεπτομέρειες, όπως τα κριτήρια ποιότητας και ούτω καθεξής θεωρούμε ότι το θέμα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το έχει εντοπίσει το Κοινοβούλιο και στο παρελθόν. Είναι ένα πρόβλημα που δεν θα φύγει από μόνο του. Υπάρχει ζήτηση για πληροφορίες και δεν είναι σαφείς οι κοινοτικοί κανόνες ως προς αυτό. Άρα, χαίρομαι που αναγνωρίζετε κι εσείς τη σημασία αντιμετώπισης του θέματος αυτού, που καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ανάγκη για ε, ακροάσεις και ούτω καθεξής. Τώρα, κάποια σχόλια. Επιτρέψτε μου για τις παρατηρήσεις που κάνετε σε ό,τι αφορά τα φυλάδια και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το φάρμακο. Όντως, στην νομοθεσία μας είχαμε ορίσει επακριβώς τι θα πρέπει να αναγράφεται στο φυλάδιο αυτό και είναι μάλιστα μακρύς ο κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να αναγράφονται. Επίσης, ε, Έχουμε εισάγει, και μάλιστα το Κοινοβούλιο το έχει ζητήσει έντονα, ε, διάφορες διατάξεις για να είναι ευανάγνωστα τα φυλάδια αυτά. Όπως είπε και ο εισηγητής, ε, ε, δεν σημαίνει ότι επειδή το γράφει ο κανονισμός, τελικά γίνονται αυτόματα ε, ευανάγνωστα τα φυλάδια αυτά. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε τη βελτίωση των φυλαδίων αυτών και να απαντήσω στην κυρία Κορτίνες ότι στην πρόταση για την φερμοεπαγρύπνηση που συζητήσαμε πριν από λίγο, εισήγαμε τις διατάξεις ακριβώς τις οποίες ζητάει. Δηλαδή ένα τμήμα, ένα κομμάτι στο φυλάδιο, αυτό που ονομάζουμε βασικές πληροφορίες ε, προϊόντος, για κάποια φάρμακα μία προειδοποίηση. Μην ε, λαμβάνετε το φάρμακο αν είστε έγκυος, για παράδειγμα, για κάποια φάρμακα. για παράδειγμα για κάποια άλλα φάρμακα κάποιες ε, οδηγίες να μην λαμβάνετε όταν πριν το φαγητό για παράδειγμα. Όλα αυτά λοιπόν περιλαμβάνονται στην ενεργειακό επαγρύπνηση. Να δώσω πληροφορίες αν θέλει κυρία Πουτέρης. Τώρα κάποια άλλα θέματα που αναφέρατε όπως για παράδειγμα η ποιότητα, η πληροφορία και η ενημέρωση στο διαδίκτυο. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό αφορά θέμα ποιότητας και μάλλον ότι είναι ποιοτική αυτή η ενημέρωση. Και υπάρχουν σχετικές διατάξεις. Προκειμένου, για παράδειγμα, να μην είναι μόνο στα αγγλικά οι πληροφορίες αυτές και ούτω καθεξή. Άρα, ω προς τους στόχους μας, δεν ε, υπάρχουν μεγάλες διαφορές από τις δικές σας προτάσεις. Ίσως χρειάζεται κάποια συζήτηση βέβαια. Να διευκρινίσω τώρα κάτι αναφορικά με την Σουηδική Προεδρία. Η Σουηδική Προεδρία θέτει ως προτεραιότητα τα, τις προτάσεις φαρμακοεπαγρύπνησης και ψευδοπυρκαφρών φαρμάκων αλλά δεν, έχουν, δεν προγραμματίζουν να δεν σχεδιάζουν να αναφερθούν σε θέματα ενημέρωσης των ασθενών. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος Ζητά και πάλι το λόγο η κυρία Προτίνης. Συγγνώμη, κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να προσθέσω, αλλά πάρα πολύ σημαντικό όμω. Αυτό που συνέβη με τη γρήπη των πτηνών και τη νέα γρήπη τώρα, την ΙΤΑ ε, 1-1, υπήρξε καλυμμένη διαφήμιση για το ταμιφλού και μου φαίνεται σκέτο σκάνδαλο. Και θα πρέπει να προειδοποιήσουμε τις κυβερνήσεις. Δηλαδή, ο κύριος Ράνσφιλτ θα τρίβει τα χέρια του. Διότι βγήκανε οι εταιρείε και ένα εμβόλιο, το πούλησαν του μοσχοπούλησαν και αγόρασαν οι κυβερνήσει γιατί τέλειω ο κόσμο θα είχε θορυβηθεί και τώρα στα σκουπίδια γιατί σιγά μην τα χρησιμοποιήσουν. Και έχουν και ονοματεπώνυμα όλα αυτά τα σκάνδαλα. Ο κύριος Ράμσφιλτ και η κλίκα του εκεί πέρα χαίρονται τώρα. Επίσης, βέβαια το, ε, το έγγραφο αυτό είναι άσχετο, αλλά εμείς στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνουμε συστημική προσέγγιση θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Το ίδιο φάρμακο ή αντίστοιχο φάρμακο να έχει την ίδια συνταγή και την ίδια αντιμετώπιση. Γιατί όμως για το ίδιο φάρμακο το ίδιο φάρμακο όταν έχει άλλο ιδιοσκεύασμα θέλει συνταγή ενώ κάποιο άλλο όχι. Τελειώνω. Για να γελάσουμε και λίγο. Στην Ισπανία βέβαια είναι θλιβερό το παράδειγμα. Το αντισυλληπτικό χάπι της επομένης ημέρας ήρθε μια μητέρα και είπε θέλω να αγοράσω ένα κουτί. Ένα κουτί ολόκληρο γιατί έχω δύο κόρες. Η μία είναι πολύ ε, και συγκρατημένη αλλά είναι θεότρελη. Και κάθε Σάββατο της δίνω προληπτικά το χάπι αυτό, της το βάζω στο φαγητό χωρίς να το ξέρει. Δηλαδή της δίνει ένα φάρμακο, μην μείνει έγκυος. Γιατί, γιατί είναι ελεύθερο το φάρμακο, κυκλοφορεί χωρίς συνταγή το ίδιο φάρμακο αλλού είναι μέση συνταγή ανάλογα με το ίδιο σκεύασμα. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε ίδια πολιτική για όλους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Χατζημαρκάκης για να απαντήσει σε αυτό το τελευταίο. Ναι. Ε, θέλω να γνωρίσω και τις δύο κόρες, καταρχάς, για να το λύσουμε το θέμα. ναι, για να με ενδιαφέρει και το θέμα έτσι από ψυχολογικής πλευράς για τα εμβόλια. Έχουν εξαιρεθεί τα εμβόλια. Με το ταμιφλού πολύ χρήσιμο αυτό που είπατε, να κάνουμε ακρόαση εδώ στο Κοινοβούλιο, τι θα γίνει, ας πούμε, αν κάποιοι που ο κύριος Σοτάδε που είπατε και εσείς έχουν πολιτικές θέσεις και ε, στέλνουν πληροφορίες μέσω από στρατιωτικά επιτελεία και κερδίζουν οι εταιρείε τους. Ε, αυτό συνέβη τώρα. Ως περήφανος Ευρωπαίος θα έψαχνα να δω αν είναι εντάξει αυτό ή όχι και με τις αμερικανικές πληροφορίες. Σας είπα προηγουμένως ότι κατευθύνονται πάρα πολλές πληροφορίες ε, ε, ε, fake πληροφορίες τις λέμε αυτό σε ωραία γερμανικά, ψευδείς δηλαδή, αλλά εξαιρούνται ήδη οι εκστρατείε εμβολιασμού. Για να γίνει ένα εμβολιασμό θα πρέπει να το εγκρίνει ο οργανισμό που είναι αρμόδιο σε κάθε κράτο, που ποικίλει αυτό. Και για τη Σουηδική Προεδρία αποφάσισε, ε, απάντησε μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί υπάρχει απόθεμα ενός φαρμάκου, Μπορεί αυτά τα θέματα να ακούγονται πολύ τεχνικά, αλλά το συγκεκριμένο είναι πολύ καλό και πολύ σημαντικό για τους ασθενείς. Χαίρομαι που έχω τόσους καλούς και ηγητές. Ο κύριος Κορέα Ντεκάμπος ήταν υπουργό και μάλιστα υγείας και έχει εργαστεί σε αυτό το θέμα από πλευρά Συμβουλίου. Αλλά κάτι που δεν καταλαβαίνουν πολύ είναι και έρχομαι και πάλι στη μητέρα μου. Οχτώ φάρμακα παίρνει η γυναίκα. Εκεί δεν είναι και τόσο μορφωμένη όπω μερικοί από εμά που καθόμαστε εδώ. Αν τα διάβαζε όλα θα τρόμαζε και δεν θα τα έπαιρνε τα φάρμακά τη. Αυτό, ναι, ξέρω. Τώρα στο Τσεντεού θα επιθυμούσατε να είχε πάρει το αντισυλληπτικό κάπτη προηγουμένως, δεν το πήρε τώρα τι να κάνουμε και με έκανε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν, δεν τα καταλαβαίνει. Και σήμερα υπάρχουν πολύ καλές μέθοδοι και πρακτικές και πολύ διαφορετικές. Σε μια εγκεκριμένη στο σελίδα θα μπορούσε κανείς να βάζει μια μικρή ταινία, ας πούμε, που να δείχνει πώς παίρνει τα φάρμακά σου και τι ενέργειες έχουν. Σήμερα έχουμε πολύ ε, καινούρια μέσα που ξεπερνάνε κατά πολύ αυτό το χαρτάκι που έχει μέσα το φάρμακο. Βάλε ένα φιλμάκι που να έχει όμως εγκριθεί προηγουμένως από το αντίστοιχο οργανισμό. Περί αυτών πρόκειται. Ε, γερνάει η κοινωνία μας, όλο και περισσότεροι άνθρωποι μπαίνουν σε αυτή την κατηγορία. Αυτό που είπε η Χριστίνα για το βάρος είναι πολύ σημαντικό και αποφασιστικό μάλιστα θα έλεγα. Πολύ συμφωνώ να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση το χρονοδιάγραμμα δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το αναβάλουμε, να το παρατείνουμε. Θα κάνουμε την ακρόαση. Ήδη έχουν γίνει αρκετέ ανταλλαγέ επιχειρημάτων και οφείλω να επενέσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι καλή η έκθεσή τη. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε πάρα πολλά. Μερικά σημεία μπορούμε να συμπληρώσουμε, όπω είπατε κι εσεί, αλλά από εκεί και πέρα. Πρέπει να πω στην Επιτροπή ότι έκανε πολύ καλή δουλειά. Βέβαια, έκανε και ένα κάρο χρόνια για να τη βγάλει αυτή τη δουλειά και τώρα επιτέλου θα πρέπει να την εφαρμόσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Και πάμε στο σημείο 9 τώρα, ψευδεπίγραφα φάρμακα. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Σαρτόρη, που περίμενε πάρα πολύ ώρα. Με υπομονή έχετε το λόγο και θα πρέπει να της αφιερώσουμε και την απαραίτητη προσοχή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με πάρα πολύ προσοχή όλη τη συζήτηση. που συνδέεται και με αυτό το θέμα, το άλλο θέμα, γιατί πρόκειται για ένα συνολικό πακέτο, πολύ σημαντικό για όλους τους πολίτες, τα φάρμακα δηλαδή. Καλό θα είναι να μπορέσουμε αυτές οι οδηγίες και οι κανονισμοί να ισχύσουν προς προστασία των πολιτών. Εγώ το θέμα μου είναι τα ψευδεπίγραφα φάρμακα. σαν είναι μια τροποποίηση της οδηγίας του 2001 του 83. 2001 του 83. Με στόχο να μην μπαίνουν στο νόμιμο κύκλωμα ψευτοφάρμακα. Επειδή υπάρχει το θέμα των ε, ενεργών συστατικών. Με βάση την δήλωση 61 του 2006, όπου ζητούσαμε να ελεγχθεί ότι η σωστή μέθοδος παραγωγής θα είναι εγγύηση υψηλής ποιότητας και για τα φάρμακα αλλά και για τις ενεργές ουσίες που βρίσκονται μέσα στα φάρμακα. Η οδηγία λοιπόν 2001 το 83 δεν προέβλεπε αυτή την υποχρέωση για τους Ευρωπαίους παραγωγούς και για τους εξωκοινωτικούς επίσης. Και αυτό ζημίωσε την υγεία του πολίτη και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας. Εμείς λέμε στην ίχνη δασιμότητα των ενεργών ουσιών και στην ανιχνευσιμότητα των, των φαρμάκων θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα σύστημα που να ισχύει για όλη την Ευρώπη. Συνήθως ε, είναι τρεις ε, ομάδες τα ψευτοφάρμακα. Το ένα αφορά την ταυτότητα, η απομίμηση, δηλαδή το προϊόν δεν περιέχει το σωστό συστατικό ή τη σωστή ποσότητα του συστατικού, το ιστορικό, έχουν φύγει από την αλυσίδα διανομής και δεν τηρούν ε, τις αυστηρές προδιαγραφές μεταφοράς και το τρίτο είναι η προέλευση. Δηλαδή εκεί που παρασκευάστηκαν είναι ο, ο τόπος είναι διαφορετικός από αυτόν που δηλώνεται στο, στο φάρμακο απάνω. Αυτές είναι οι τρεις ομάδες απατών ή απομίμησης. Ξέρουμε ότι με βάση τον ΠΟΗ το 1% των φαρμάκων στις γεωμικές χώρες είναι ψευτοφάρμακο από μίμηση. Δεν είναι λίγο. Μιλάμε για φάρμακα. Μιλάμε για φάρμακα τα οποία κάνουν καλά τον πολίτη. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι το ποσοστό αυτό αυξάνει κατά 20% κάθε χρόνο. Πέρα λοιπόν από το θέμα προβλήματος της υγείας των πολιτών, Μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο κουτιά φαρμάκων από μιμήσεις που κάθε χρόνο μπαίνουν στην αγορά της Ένωσης. Έχουμε και ένα πρόβλημα εσωτερικής αγοράς. Όταν μιλάμε για τις φαρμακοβιομηχανίες, μιλάμε περίπου για χίλιους παραγωγούς γενικών φαρμάκων και άλλους χίλιους άλλου είδους φαρμάκων. 650.000 απασχολούμενοι 1.500 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 17% των ευρωπαϊκών δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη. Και γι' αυτό, επειδή τα νούμερα αυτά είναι μεγάλα για τη βιομηχανία, το ποσοστό της φαρμακοβιομηχανίας, ζήτησα συνεργασία, ενισχυμένη συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, γιατί αφορά και την υγεία των πολιτών, αλλά αφορά και ένα σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Σήμερα το 31% των φαρμάκων μαϊμού προέρχεται από την Ινδία, το 31% από τα Αραβικά Εμμυράτα και περίπου 25% από την Κίνα. Οι προτάσεις της Κομισιόν στις οποίες θα προσθέσουμε και εμείς ορισμένα σχόλια είναι οι εξή. Πρώτον, πρέπει η Ευρώπη να προωθήσει σε διεθνή όργανα όπως στον ΠΟΕ και λοιπά ή στην τον κόσμο οργάνωση, οργανισμό υγείας ένα πλάνο να καταπολεμηθεί αυτή η παρουσία αυτών των ψευτοφαρμάκων γιατί δεν εκτιμούν τον κίνδυνο όλοι σε παγκόσμιο επίπεδο με τον ίδιο τρόπο. Το δεύτερο, για όσα ισχύει η νομοθεσία, και μέχρι στιγμής μιλούσαμε για καλές μεθόδους, αφορούσε τους κατασκευαστές, παρασκευαστές και τους διανομείς. Υπάρχει μια καλή μέθοδος παραγωγής και μια καλή μέθοδος διανομής του φαρμάκου. αλλά ειδικά για τη διανομή πολλές φορές συνδέεται και με άλλα θέματα που δεν τα έχουμε αντιμετωπίσει και συζητήσει. Οπότε λείπει ένα νέο τρίτο στοιχείο. Υπάρχουν και άλλα οντότητες πέρα από τους παραγωγούς και τους διανομής. Αυτά τα διαφορετικά άτομα ή επιχειρήσεις μπορεί να είναι μεσολαβητέ, κάποιο που αγοράζει για λογαριασμό ενός τρίτου μια παρτίδα φαρμάκων από μια χώρα και τα πουλάνε σε άλλη. Οι έμποροι που αγοράζουν για δικό του λογαριασμό ένα φάρμακο και μετά τα πουλάνε. Αυτές οι νέες κατηγορίες ενδιαμέσων που έχουν εμφανιστεί στην αγορά πρέπει και αυτές να ρυθμίζονται. Τρίτο, ποιος εγγυάται την πιστοποίηση των σωστών μεθόδων παραγωγής, άρα την μη απομίμηση. Ό,τι προέρχεται από το εξωτερικό της Ένωσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των μονάδων παραγωγής από τις εθνικές αρχές της Ένωσης. Και δεν μιλάμε μόνο για γενικά φάρμακα, αυτό ισχύει και για τις, ε, ε, τα ενεργά συστατικά. Διότι εισάγουμε το πιο μεγάλο ποσοστό των ενεργών ουσιών που χρησιμοποιούμε στα φάρμακά μας. Ένα ασθενέ σημείο ότι έχουμε, είναι ότι έχουμε κατά νου δύο λίστες Στη μία είναι τα κράτη όπου υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο παρόμοιο ή και καλύτερο από το ευρωπαϊκό. Αλλά για να το ελέγξουμε αυτό μας χρειάζονται τρία χρόνια. Εγώ θα έλεγα να μειωθεί αυτό το διάστημα. Όχι τρία χρόνια. Στο δεύτερο μέρος δεν υπάρχει λίστα θα πρέπει ή οι εθνικές αρχές ή κάποιος άλλος να μπορεί να κάνει αυτή την πιστοποίηση. Τέλος, η οι εθνικε αρχες η καποιο αλλο να μπορει να κανει αυτη την πιστοποιηση τελος η χνηλασιμοτητα του προϊόντο. Αυτό είναι απολύτως αναγκαία για να κατοπρομηθεί η απομίμηση των φαρμάκων. Μόνο δηλαδή αν καταλάβουμε πού γίνονται και τι διαδρομή ακολούθησαν τα συστατικά ή το φάρμακο, μόνο τότε θα μπορούμε να έχουμε ένα πιο σωστό έλεγχο. Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο πρόβλημα, οι κυρώσει. Σήμερα δεν, δεν μετράνε οι κυρώσει αυτές. Αν κάποιος δράει εγκληματικά, αν κυκλοφορεί ας πούμε πλαστά φάρμακα, Εκεί είναι λίγο πιο αυστηρές οι, κυρώσει. Αλλά δεν είναι ισοδύναμες από χώρα σε χώρα. Μετά υπάρχει ο κίνδυνος, η πόλη στο φαρμάκο μέσω του ίντερνετ βοηθάει στο να πουλιώνται πλαστά φάρμακα. πιθανώς να μην είμαστε σε θέση με αυτή την αλλαγή της οδηγίας να λάβουμε υπόψη όλα όσα έχουν σχέση με τις πωλήσει μέσω ίντερνετ. Τελευταίο. Ο χρόνος που προβλέπεται για να ισχύσει η οδηγία 18 μέχρι 48 μήνες αν μπορούσαμε να το μειώσουμε λίγο επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό θα ήταν προτιμότερο 18 μέχρι 36 μήνες τελειώνω με κάτι άλλο είχαμε πολύ, μερικά πολύ σοβαρά κρούσματα πρόσφατα όπου πέθαναν άνθρωποι όχι σε σχέση με την παραποίηση του φαρμάκου αλλά οι οδηγίες ήταν τελείως λάθος. Μεγάλη ζημιά είχαμε θανάτους σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα στις αναλυσσόμενες χώρες. Πρέπει και γι' αυτό να υπάρχουν οι κανόνες. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ε τώρα οι σκιώδεις ηγητέ, η σοσιαλίστρια κυρία Μέρκης ε, είναι ε, ε, από απούσα και σε καταπληκτικά γερμανικά μου φέρνει ένα σημείωμα που λέει ότι την αντικαθιστά ο κύριος Κορέντε Κάμπος, ο οποίος είναι τιμοπόλεμος σε όλα τα μέτωπα από ό,τι βλέπω. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα γερμανικά μου δεν είναι καλά και θα πω αγγλικά αν με επιτρέπετε. Ε, λόγω ανελημμένων υποχρέωσεων στι κάτω χώρε, δυστυχώ η Judith η ε, σκιώδης κολλή τη σήμερα και μου ζήτησε να τα πω εγώ εξ ονόματό τη. Θα πρέπει καταρχάς να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δουλειά τη. Ε, και τη λεπτομερή πρόταση. Σύντομα θα σας πω τι λέει η σκιώδη συζηγήτρια για την πρόταση που αφορά την πρόταση ε, για να μην μπαίνουν ψευδεπίγραφα φάρμακα στην κυκλοφορία στην αγορά. Η ασφάλεια και η υγεία του στενούς είναι πάντα το πρώτο μας μέλημα και θα πρέπει το γενικό συμφέρον του καταναλωτού να είναι πάντα στο μυαλό μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει μόνο το άρθρο 95 των συνδικών σε σχέση με αυτό. Μα θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως θα πρέπει να βάλουμε στην οδηγία και άλλα άρθρα. Παράδειγμα, 152 για τη δημόσια υγεία. Δεύτερον, πριν αρχίσουμε τη συζήτηση επί της ουσίας για το θέμα αυτό, θα πρέπει να ορίσουμε τι είναι τα πλαστά φάρμακα. Διεθνής ορισμός ε, ευρέως παραδοκτός θα ήταν ευχής έργο, αλλά δυστυχώς απουσία ε, διεθνούς ε, ορισμού η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πρόοδο. Μετά το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας είναι για φάρμακα μόνο υπογρατικής συνταγογράφησης. Ωστόσο θα πρέπει να δούμε τι είδους φάρμακα είναι αυτά και τι φαρμακευτικά σκευάσματα θα μπουν. Παράδειγμα, τι κάνουμε με τα κοινόχρηστης ονομασίας και αν θα πρέπει να μπαίνουν και τα, οι πρώτες ύλε στην οδηγία. Γιατί δεν είναι αρκετά σαφής η εισηγήτρια, λέει η κυρία Μέρκης. Μετά, τα φάρμακα που κυκλοφορούν στα κράτη-μέλη, θέλουμε να είμαστε πιο διαφανείς στην προσφορά μας, θα πρέπει να ξέρουμε πώς πουλάμε τα φάρμακα. Έτσι θα βελτιωθεί η διαφάνεια. Πέμπτον, θα πρέπει να τονίσουμε το εξής. Πώς δεν θα υπάρξουν διαρροές για να μπαίνουν στη νόμιμη αγορά και στην αλυσίδα παραποιημένα φράγματα, ε, φάρμακα συγγνώμη, και ε, μην έχουμε προβλήματα στην υγεία των ασθενών. Βεβαίως καλύτερη ένδειξη, ε, αλλά θα πρέπει να έχουμε και στοιχεία ασφάλειας διαφόρων κατηγοριών κινδύνων και αναλογικά, γιατί το κόστος για τον καταναλωτή θα πρέπει να παραμείνει όσο γίνεται πιο χαμηλό. Στη συνέχεια, είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια των επόμενων συζητήσεων να πούμε ποιος θα είναι αρμόδιος για το σύστημα εχνηλασιμότητας και τη βάση δεδομένων. Να σεβόμαστε και την ιδιωτική ζωή και το απόρριτο της βιομηχανίας των ιδιωτικών εταιριών. Θα πρέπει λοιπόν η βάση να είναι τελείως ανεξάρτητη. Το βασικό θέμα εδώ δεν είναι η ενημέρωση, αλλά ο κίνδυνος και η ασφάλεια. Τέλος, και είναι σημαντικό αυτό, πρέπει να πούμε ότι το διαδίκτυο είναι από τις βασικές πηγές παραποιημένων φαρμάκων. Τα περισσότερα ψευδεπίθερα κυκλοφορούν από το ίντερνετ. Πολύ μεγάλες ποσότητες, πάνω από το μισό, 62% των φαρμάκων που κυκλοφορούν ε, και απολούνται στο ίντερνετ μπορεί να είναι ψευδεπίγραφα. Θα πρέπει να έχουμε αυστηρότερους κοινούς κανόνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Χατζημαρκάκης παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη συνάδελφο γιατί και αυτή τη φορά έκανε πάρα πολλές ε, σημαντικές και σωστές παρατηρήσει. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το διαδίκτυο, ότι το διαδίκτυο αποτελεί τη βασική πηγή για τα ψευδεφύγραφα φάρμακα και υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες έχουν καταδείξει το σχετικό και μάλιστα ο μιλάει, η ΠΟΕ μιλάει για 50% σχετική μελέτη η Γερμανικού Ιδρύματος μιλάει για 80% ποσοστό ε, ψευδεπίγραφων φαρμάκων στο διαδίκτυο. Λοιπόν, θα πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης του προβλήματος αυτός. Θα μπορούσε να υπάρχει ένας ε, κατάλογος, για παράδειγμα, με τα πιστοποιημένα φαρμακεία μέσω του διαδικτύου, για να παίρνει κανείς πιστοποιημένα ε, προϊόντα. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν προηγηθεί μια μεγάλη εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του πολίτη κάποια προϊόντα lifestyle, ξέρω εγώ, από την ε, Ανατολική Ασία, ε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ε, είναι πρωτότυπο το φάρμακο, το προϊόν. Το θέμα του κόστους τώρα. Το θέμα της επισήμανσης το οποίο αναφέρει η Κομισιόν έχει να κάνει με το κόστος. Και χαίρομαι που πριν από κάποιες εβδομάδες διοργανώθηκε μια εκδήλωση και συμμετείχε και η συγγήτρια και πολλά στοιχεία τα συμπεριέλαβε. Και αυτό κατέδειξε για μία φορά ακόμα πώς μικρές επιχειρήσεις ε, του φαρμακευτικού κλάδου επιβαρύνονται με τεράστιο μαζικό κόστος και αυτό να το λάβουμε υπόψη κατά την υποβολή της πρότασης αυτής και θα πρέπει να ανάλογα προς ανάλογη κατεύθυνση να κατευθυνθεί και η τεχνολογία. Τελευταίο σημείο. Όντως, δεν συμπεριλαμβάνονται οι πράκτορες. Θα πρέπει και αυτοί να συμπεριληφθούν. Θα πρέπει να υπάρχει και ένας σαφής κώδικα σε περίπτωση ε, εισαγωγής φαρμάκων στην εμπόριο και των σχετικών κυρώσεων. Ωστόσο, τέτοια στοιχεία περιλαμβάνονται και από την πρόταση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής πιο πολύ θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε ως επόπτες, όχι μόνο ως άτομα που είναι υπεύθυνα για την παραβίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή... Α, συγγνώμη, η... Μεγάλο μου λάθος. Συγχωρέστε με. Δική σας σειρά. Ναι, όχι, όχι. Συγγνώμη, Πρόεδρε, δεν ήθελα να πάρω το λόγο, αλλά σας ευχαριστώ Θα ήθελα και εγώ να διευκρινίσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να συζητηθεί η έκταση αυτή και σε μια άλλη επιτροπή. Να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Τα σημεία που έθιξε η συγγήτρια και ο συνάδελφος Κάμπος, τα σημεία λοιπόν που αναπτύχθηκαν ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη σημασία και ε, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι σε συνεργασία με τους συναδέλφους ε, θα καταφέρουμε πολλά και θεωρώ ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σημειώσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα πρόοδο. Δεν ξέρω είναι δυνατή ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα αυτό για να διατυπώσουμε και κάποιες παραπάνω ιδέες και να υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες. για την έκθεση στις 3 Δεκεμβρίου. Προκειμένου και εμείς να εξετάσουμε στην τροπολογία σε όλα αυτά τα θέματα. Μάλιστα, νομίζω ότι είναι καλή προσφορά ε, για τους συναδέλφους εδώ στην Επιτροπή. Και να δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Σάντσες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you, Chair, and, um, Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και για την ενίσχυσή σας, την υποστήριξή σας για την γρήγορη ανάληψη δράση για να καταπολεμήσουμε την ε, παραποίηση των φαρμάκων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ε, πολλά συγκεκριμένα στοιχεία ακούσαμε. Να προσπαθήσω να σας απαντήσω. Αλλά θα επικεντρωθώ σε δύο-τρία βασικά θέματα. Το θέμα των ορισμών. Το έθιξε η κυρία Σαρτόρη και ο κύριος Κάμπους να σας ε, διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συμμετέχει στους διεθνείς, στις διεθνείς συζητήσεις για να καταλήξουμε σε κοινούς ορισμούς. Τελικά το εγχείρημα αποδεικνύεται πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει σαφής ορισμός στο κείμενο, αλλά από τον τίτλο της πρότασης και από τη χρήση των ίδιων κειμένων της άλλες θα προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε το τι ακριβώς αντιμετωπίζουμε στο σημείο αυτό. Όπως είπε η κυρία Σερτόρη, πρόκειται για φάρμακα τα οποία έχουν παραπλαστογραφηθεί ε, ως προς την πηγή τους, την ιστορία τους, προϊόντα τα οποία δεν είναι αυτό που ισχυρίζονται ότι είναι. Και για σκοπούς δημόσιας υγείας, ανεξάρτητα από θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, μας απασχολεί το θέμα αυτό. Το, λέω αυτό γιατί υπάρχουν και ορισμοί στο κοινωτικό δίκαιο ε, παραποιημένων προϊόντων ε, οι οποίοι σχετίζονται με πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Και εδώ μας απασχολούν φυσικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά προέχει η υγεία του ασθενή, γιατί το προϊόν δεν περιέχει αυτά που λέει ότι έχει. Γι' αυτό λοιπόν για μας είναι σημαντικό να διατηρηθεί αυτή η έννοια της ε, πλαστογράφησης, της ιστορίας, της πηγής και της σύστασης. Κάτι πολύ βασικό για θέματα ιχνηλασιμότητας και για να καθοριστεί το τι θα προταθεί είναι να ισορροπήσουμε την προστασία της δημόσιας υγείας και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε για να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά που είναι αρκετά υψηλοί αν εισαχθούν και διατάξεις αναφορικά με την ασφάλεια. παρέχουμε σχετική επιχειρηματολογικία στην μελέτη αντικτύπου και σας ζητώ να το λάβετε αυτό υπόψη, όπως ανέφερε και ο κύριος Χατζημαρκάκης. Μια άλλη πτυχή η οποία αναφέρθηκε προφανώς ε, προήλθε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα το πώς θα ε, αντιμετωπίσουμε το θέμα της εισαγωγής δραστικών ουσιών. Επειδή πολλά από τα φάρμακα περιέχουν δραστικές ουσίες που έχουν εισηχθεί από τρίτες χώρες βάλαμε κάποιες διατάξεις πολύ καινοτόμες στην ε, νομοθεσία μας και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε, όπως είπε και η συγγήτρια, ότι οι καλές πρακτικές των παραγωγών και στο θέμα της διανομής θα γίνουν σεβαστές. Ωστόσο, να κάνω ένα σχόλιο για την πρόταση αυτή. Να πω ότι μπορεί να χρειαστεί να μας ε, διαβεβαιώσει η αρμόδια αρχή μας ότι έχει εκτελέσει ελέγχους. Περίπου 20.000 σχέδια υπάρχουν ε, για τις δραστικές αυτές ουσίες και αν κοιτάξουμε όλες τις εκθέσεις γίνονται περίπου 60 επιθεωρήσεις ανά έτος. Άρα θέλουμε να βρούμε λύσεις οι οποίες να είναι και εφαρμόσιμες στην πρόταση, προκειμένου να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία, να διασφαλίσουμε την καλή παραγωγή και τις καλές ε, πρακτικές ε, διανομής με συστηματικές ε, επιθεωρήσεις, αλλά να μην αντιμετωπίζουμε τελικά και ένα πρόβλημα εφαρμογής. Λοιπόν, να το έχουμε και αυτό υπόψη. Επίσης αναφέρεται θέματα ως προς το πεδίο εφαρμογής, και για άλλα είδη ουσιών, όπως τα έκδοχα και για ε, ενδεχόμενη επέκταση του πεδίου εφαρμογή ε, πέρα από τις δραστικές ουσίες θα πρέπει να βασιστούμε ε, σε αξιολόγηση κινδύνου. Είναι πιο χαμηλός ο κίνδυνος, γιατί έχει γίνει μια μελέτη δεκτή που πρόσφατα από ότι για τις δραστικές ουσίες και δεν νομίζω ότι θα μπορούν να ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι κανόνες και για τα έκδοχα. Ένα τελευταίο τώρα σημείο, το οποίο θίξετε επανειλημμένα, το διαδίκτυο. Γενικά συμφωνούμε με αυτό που είπε η κυρία Σαρτόρη, ότι μπορεί να μην ε, καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε το θέμα του διαδικτύου σε αυτή την πρόταση, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι θα πρέπει να ρυθμίσουμε και τη λιανική πώληση των φαρμάκων, το οποίο δεν εντάσσεται στο σύστημά μας σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν και δεν το καλύψαμε στην πρότασή μας, γιατί αυτό ε, να πόκεται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αλλά όντω υπάρχει δυνατότητα να επιληθούν κάποιες πτυχές του προβλήματος. Θα περιοριστώ γιατί βλέπω ότι περνάει και η ώρα και έχει περάσει 6.30. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτό που είπατε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους τέσσερις αναπομείναντες βουλευτές, τους γραμματείς, τους διερμηνείς ιδιαίτερα που κάνουν υπερορίες και τους προσκεκλημένους μας. Ε, καλό σας βράδυ και καλή επάνωδο.